και η άποψη της μειοψηφίας συγκεκριμένα των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων και της Γκουε. Έτσι είναι. Τώρα φωνάζω και με πιάνω ο μου. Λοιπόν, Κορίν, είχε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξ' του ΕΛΚ θεωρούμε δεδομένης της κρίσης και της κατάστασης στην Ελλάδα πως είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να ψηφίσει επί της θέσης μας για το που βρισκόμαστε στο πακέτο διακυβέρνησης και σε μεγάλο βαθμό και χαιρόμαστε γι' αυτό ε, συμφωνούμε νομίζω με το Συμβούλιο ε, χάρη στην δουλειά που έγινε από την ομάδα Συμβουλίου και Κομισιόν και θα ήθελα να αναφέρω εδώ πέρα τον Άντρες Κάρμαν, δεν ξέρω αν είναι στην αίθουσα, εδώ είναι. Θα ήθελα ιδιαίτερα τον Άντρες Κάρμαν να ευχαριστήσω γιατί επέδειξε μεγάλη υπομονή και αποφασιστικότητα και ισχυρά επιχειρήματα στην ε, συζήτηση αυτή για να φτάσουμε εδώ και αυτό δεν ήταν εύκολο και είναι ε, εύκολο βεβαίως ε, να κατηγορεί κανείς και να λέει πως όλα λάθη Αυτό το οποίο κάνατε όμως ήταν πάντα σωστά και επιτύχαμε πέμπτη πρωί στις 3 η ώρα να έχουμε ένα αποτέλεσμα μετά από 12 ώρες διαπραγμάτευσης. Ε, εσείς ήσασταν 24 ώρες το πόδι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πραγματικά προχωρήσαμε πολύ μακριά. Θέλουμε λοιπόν να πάμε σε ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα για να ξεκαθαρίσει η θέση του Συμβουλίου, αλλιώς θα ευλογήσει αν θέλετε τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ το Συμβούλιο και πάπαλα τελείωσε. Θα είναι εκτός το Κοινοβούλιο και δεν νομίζω βεβαίως να σας προξενήσει η έκπληξη πως ε, είχαμε σοβαρά προβλήματα με κάποια από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Τρίτης και άρα διακυβεύεται η πλειοψηφία στήριξης του πακέτου στο Κοινοβούλιο και αυτό δεν το θέλουμε. Και βλέποντας τις εξελίξεις στο Συμβούλιο και εδώ πέρα το είπε και ο Ζαν Πολκουζές πρέπει να θυμόμαστε το 2003-2005 τι έγινε. Πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά οι αποφάσεις και να είναι αποτελεσματική η διαδικασία σε Συμβούλιο και Κομισιόν. Γι' αυτό θέλει το Κοινοβούλιο να επιμείνει η αρχή της διαδικασίας κυρώσεων, μιλάμε για κυρώσεις, να υπόκειται σε αντιστραμμένη ειδική πλειοψηφία. Δεύτερον, που θα ήθελα να αναφέρω, είναι πως μετά από μακροσκελής πραγματεύσεις μεταξύ των ε, διαφορετικών ε, πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο βρήκαμε μια κοινή γραμμή σε σχέση με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και την έκθεση Ελίζα Φερέρα για συμμετρία και ασυμμετρία και ποια είναι η προσέγγιση όταν μιλάμε για μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ήταν μια δύσκολη ισορροπία και χάρη στην πρόοδο ε, που επετεύχθη τρίτη βράδυ νομίζω πως καταλήξαμε σε μια γραμμή που θεωρούμε πως πρέπει να δεχτεί το Συμβούλιο. Δηλαδή συμμετρική όπου δει. Και αυτό νομίζω έγινε δεκτό και από το ΕΚΟΦΗΝ και είναι κάτι σημαντικό το οποίο θέλει να κρατήσει το Κοινοβούλιο. Οπότε εγώ εξ ονόματος του ΕΛΚ θέλω να πω αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Μπόλς. Δηλαδή να πάμε στην ψηφοφορία να ε, Τεχθεί σε ψηφοφορία το αποτέλεσμα της ε, τρίτης πρωινή ε, συν μια τροπολογία επί της αντίστροφης ειδικής ε, πλειοψηφία, το οποίο επιμένει το Κοινοβούλιο. Νομίζω πω είναι υπεύθυνη αυτή η στάση και ξεκαθαρίζουμε και στον εξωκόσμο το ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Αν και γνωρίζω πως ειδικά όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας υπάρχουν ακόμα αποκλίνουσες απόψεις εντός του Κοινοβουλίου αλλά για το ΕΛΚ υγιή δημόσια οικονομικά. Το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θέμα κλειδί και άρα μπορούμε να στηρίξουμε το πακέτο όσο έχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ούντο. Κυρία Πρόεδρε, η ομάδα μας πάντα έλεγε πως χρειαζόμαστε σταθερά δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό είμαστε πάντα στη διάθεσή σας ε, για ένα καλό πακέτο και για διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο αλλά θα πρέπει να το μπορούμε να το επιτύχουμε. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με ποινές. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική ισορροπημένη της ανάπτυξης και να προστατεύουμε τον πυρήνα τον αναπτυξιακό και να έχουμε και τον πυρήνα και την ε, πτυχή της ε, βιωσιμότητας και της δικαιοσύνης και των στόχων του 2020. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Βόρτμαν Κόλ πηγαίνει πολύ παραπέρα επιβάλλει μια λογική λιτότητα με εξαιρετικά μικρές ε, πλειοψηφίες χωρίς να μπορεί να ε, ενημερωθεί όλο το κοινοβούλιο για το ποιο ήταν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Είναι προβληματικό αυτό, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας δε. Ειδικά στην περίπτωση στην, οποία βρίσκεται, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη, δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα διάσωσης, δεν επιτρέπεται να πούμε πως ε, θα κάνουμε τώρα τα τάγματα σκαπανέων, τιμωρίας εάν θέλετε και μετά θα δούμε ποια θα είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Όχι. Για λόγους λοιπόν διαφάνειας είμαστε κατά αυτής της διαδικασίας. Νομίζω πως ε, θα ήταν απλούστερο να πάμε τον Ιούλιο να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις προτάσεις και μετά να καταλήξουμε σε μια νέα συνένεση. Σας παρακαλώ ακόμη μια φορά εξ ονόματος της ομάδας μου να ε, προσπαθήσουμε να έχουμε ένα συμβασμό το, στον οποίο θα συμφωνήσει ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς βεβαίως η Βρετανή Συντηρητική και το ECR είναι κατά. Το ΕΛΚ ε, απάντησε αρνητικά. Όπως είπε δηλαδή ο Ζαν Πολγκοσές δεν ξέρει καν περί τίνος πρόκειται. Αναμένουμε απάντηση από την Άλντε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της ομάδας στην αίθουσα. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια απάντηση. Για εμένα είναι σημαντικά αυτά για την ε, πολιτική μας ε, συμπεριφορά. Θεωρώ ακόμη μια φορά αν πάμε στον Ιούλιο και έχουμε ευρύτερη πλειοψηφία στο ε, Κοινοβούλιο αντί για μικρές μικρές πλειοψηφίες για να ψηφίσουμε κάτι το οποίο συμφωνήθηκε τρεις η ώρα το πρωί, νομίζω θα είναι καλύτερο. Και παρακαλώ να στηρίξετε την πρότασή μου. Ευχαριστώ, η Σίλβη. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους εργάστηκαν κοπιαστικά σε αυτό το ντοσιέ για μήνες ολόκληρους, πολύ δύσκολο και μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα άντεξε η ομάδα των διαπραγματευτών και των εισηγητών και η, ε, η γραμματεία μας βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διατύπωση και όλοι ρεν ε, παρόλο που υπέστη τεράστιες πιέσεις και είχε πολλή δουλειά με την Ελλάδα, ήρθε παρόλα αυτά και στη δική μας συνεδρίαση. Έχω δύο παρατηρήσεις επί της ε, διαδικασία και μία επί τη Ό,τι αφορά το πώ αντιλαμβάνεται το Συμβούλιο τη Συνδιαλλαγή, θα ήθελα να εκφράσω την τεράστια απογοήτευσή μου. Μιλάμε για το Συμβούλιο που απαρτίζεται από κυβερνήσει που ίδιε ήθελαν να ε, να συμφωνήσουν και να ακυρώσουν τη συνθήκη της Λισαβόνας που μας έδωσε τέτοιες εξουσίες. Αφού τη στιγμή λοιπόν που ήθελαν αυτή την συνθήκη, γιατί δεν την σέβονται. Γιατί συναπόφαση δεν είναι να αποφασίσει το Συμβούλιο και να καλοπίζει κάπως την απόφαση το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει αυτό το μήνυμα να το αντιληφθεί το Συμβούλιο. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς τις δυσκολίες και θα τις λάβουμε υπόψη, αλλά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες ε, έχοντας κατά νου το γενικό κοινοτικό συμφέρον και όχι τα εθνικά συμφέροντα ή τα συμφέροντα εθνικής πολιτικής. Πολύ απογοητευτικά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Όχι μόνο για το θέμα της αντιστραμμένης ειδική πλειοψηφίας όπου δεν σημειώσαμε πρόοδο, ε, είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια διάλυσης ε, του πακέτου των μακροοικονομικών εργαλείων. Πολύ δυσάρεστο αυτό, πολύ σοβαρό και φαίνεται ότι όχι μόνο είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν ουσιαστικά το σύμφωνο σταθερότητα, αυτό που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο είναι ότι έχουν επιφυλάξει να εφαρμόσουν και το σύμφωνο Ευρώπη-ΣΥΝ που πρόσφατα σχεδίασαν. Γιατί το να εφαρμόσουμε τη συμμετρία, τον κοινό έλεγχο για όσου έχουν το κοινό νόμισμα, δεν είναι κάτι που εφήβρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μια αναγκαιότητα. Ω προ την ουσία τώρα. Οι φιλελεύθεροι θα συμφωνήσουν με την πρόταση να ψηφίσουμε με τη ΒΕΜΤΗ, αφήνοντας μια πόρτα ανοιχτή όμως. Δεν θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση με το Συμβούλιο και θα συνεχιστεί η συζήτηση και μεταξύ μας φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει όμως και ε, ένα θέμα χρονοδιαγράμματος που είναι αποφασιστικό. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πέμπτης και Παρασκευής και αν οι κρατών και κυβερνήσεων επιληφθούν του θέματος και λάβουν υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω να, η γνώμη αυτή να είναι ενιαία, γιατί αν δεν την εκφράσουμε, τότε όλες οι ομάδες θα πρέπει να καθίσουν κάτω και να εκπονήσουν νέα θέση. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό αφορά τα ευρωομόλογα. Δέχτηκα στο κείμενό μου πολλές παραχωρήσεις προς την πλευρά του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, αφαιρέσαμε κάποιες μνήες που για μας ήταν πολύ σημαντικές. Κάναμε παραχωρήσεις προς το Συμβούλιο, αλλά το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε είτε μία απερίφραστη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε αν δεν έρθει η Επιτροπή να κάνει δήλωση, να συμπεριληφθεί στο κείμενο η δήλωση αυτή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, πέραν τη δική μου έκθεση, έγιναν τεράστιε προσπάθειε, άκουνα έργο και για τα νέα εργαλεία από τη Λίζα Φερέρα, τεράστιο έργο έγινε προετοιμάζοντα την έκθεση πρωτοβουλίας της Περβάνς για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οι κυρώσει για την απάτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ε, προσέφερε μεγάλη υπεραξία. Δεν θα πρέπει να τα εγκαταλείψουμε όλα. Και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό διάλογο, όταν υπάρχει ε, άλλη εξάρτηση, είναι σημαντικό να μιλούν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη. Ο Φιλίπ, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι οι πράσινοι είμαστε υπέρμαχοι μιας αυστηρής οικονομικής διακυβέρνησης, αποφασιστικής. Θα πρέπει να πληρεί όμως αυτή τρία κριτήρια. Να είναι αποτελεσματική φυσικά αυτή η διακυβέρνηση, προφανώς, να είναι και βιώσιμη, να χαρακτηρίζεται από μια ειφορία και τρίτον, να είναι και δίκαιη αυτή η οικονομική διακυβέρνηση. Εκεί πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο πακέτο υστερεί. Γι' αυτό ε, θέλουμε να το τροποποιήσουμε κάπως, γιατί έχει με κάποια καλά σημεία, αλλά και κάποια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ανέφερα. Σε ό,τι αφορά το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η έκθεση Βόρτμαν Κόλ ε, θα καταψηφιστεί από τους πράσινους. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία. Ο πρώτος ε, λοιπόν κρίκο, είναι ότι δεν έχουμε αυστηρή ε, πειθαρχία όχι μόνο για τι δημόσιε δαπάνε, αλλά δεν έχουμε αυστηρή πειθαρχία ούτε για τι επενδύσει ούτε για την καταπολέμηση τη φτώχεια, των κλιματικών αλλαγών, την εξασφάλιση τη απασχόληση κτλ. Δυστυχώ δεν έχουμε αυτή την πειθαρχία που χρειαζόμασταν. Έχουμε την Ευρώπη του 2020, αλλά ε, κανένα δεν ενδιαφέρεται πια. Έχει γίνει γελίο το θέμα της στρατηγικής του 2020. Θέλουμε πειθαρχία, δεσμευτική πειθαρχία και για την Ευρώπη του 2020. Αν δεν μπει αυτό στην έκθεση, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με την έκθεση Βόρτμαν Call. Δεύτερον, δεν μπορούμε να έχουμε μία δημοσιονομική δημοσιότητα αν δεν έχουμε εξορόπιση εσόδων και εξόδων. Και σε ό,τι αφορά τα έσοδα και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρώτα απ' όλα ήταν κατά οποιασδήποτε προόδου εγώ υποστήριξα το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη ω πρώτο βήμα. Αν ήξερα όμω ότι σε λίγο θα είχαμε και το πακέτο τη φορολογία, αλλά δυστυχώ πόρο απέχουμε από αυτό, είναι σαν να μην υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Γι' αυτό και το συνολικό πακέτο, κατά τη γνώμη μα, δεν χαρακτηρίζεται από ισορροπία. Άλλο τώρα το θέμα τη μακροοικονομική εποπτείας. Εδώ έχουμε κάποια νέα στοιχεία, ένα νέο πλαίσιο. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που προκάλεσαν την κρίση στην Ισπανία, Ιρλανδία και αλλού. Και από αυτή την άποψη έχουμε αισθητή πρόοδο. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά αυτό που είπα και πριν και κλεισμένο των θυρών. Ένα τέτοιο πακέτο θα είναι αξιόπιστο μόνο αν η μακροοικονομική εποπτεία είναι αμφίδρομη και φυσικά όπου δει, όπου έχει νόημα να εξετάζουμε και τις χώρες που έχουν έλλειμμα και αυτές που έχουν πλεόνασμα. Αυτό είναι το θέμα το περίφημο της συμμετρίας. Το Συμβούλιο α, επίμονα και ξεροκέφαλα αρνείται κάτι τέτοιο και γνωρίζουμε γιατί. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για το σημείο αυτό και μάλιστα μερικοί θα ήθελαν περισσότερη φιλοδοξία, άλλοι λιγότερη Πάντως η συμφωνία είναι καλή και αν επιμείνουμε σε αυτή τη συμφωνία θα ψηφίσουμε υπέρ του πακέτου για τη μακροοικονομική εποπτεία. Τέλος, η Ρίκη Φόρντ ε, για τα δημοσιονομικά πλαίσια ήταν πολύ καλό, γι' αυτό και θα υποστηρίξουμε και αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε επαγγελματικούς τρόπους κατάρτισης των προϋπολογισμών. Και τέλος, μία παρατήρηση. Πολλά υπόθηκαν ε, για το Παρίσι και το Βερολίνο τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, εγώ κατάγομαι από μια μικρή χώρα, αλλά γνωρίζω ότι τίποτα μεγάλο δεν έχει γίνει στην Ευρώπη χωρίς ε, μια ισχυρή και αποφασισμένη ηγεσία και συνεργασία Παρισιού και Βερολίνου, Γαλλίας και Γερμανίας. Είναι οι μεγαλύτερες χώρες και οι μεγαλύτερες κοινωνίες στην Ευρώπη, πιο ισχυρέ οικονομίες. Yeah. Θα πρέπει να δείξουν ηγετικό ρόλο έτσι να χαράξουν το δρόμο για ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Τελικά τι κάναμε, μια πολύ μετριοπαθή η συμφωνία που υπαναχωρεί. Ε, ας αποτρέψουμε την αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία και εγώ θα σας βοηθήσω ε, να αποφύγουμε τη συμμετρία. Αυτό σημαίνει ηγεσία και όχι η απόφαση που έλαβαν Παρίσι και Βερολίνο που αποβαίνει σβάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ελίσσα και ο Κάρλ περιμένουν να λάβουν το λόγο που είναι και αυτοί οι συγγητές. Ακούσαμε έναν ομιλητή από κάθε ομάδα, αλλά έχουμε και την Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Βερμούδας που προβλεπόταν να ξεκινήσουμε ανταλλαγή μαζί της στις 10.30 και έχουμε και ανταλλαγή απόψε με το Συμβούλιο αργότερα. Παρακαλώ λοιπόν, για να μην περιμένει ο Πρωθυπουργό, να είστε σύντομοι. Θα ακούσουμε και τον κύριο Φαγιό, που είναι εισηγητή, αλλά κανέναν άλλον πέραν των εισηγητών. Εκτό και να έρθει και άλλο εισηγητή. Αλλά μόνο θα ακούσουμε όχι άλλου ομιλητέ. Η Ελίζα, ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικότατη. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τον Ούτο Βούλμαν για το πόσο ανεπαρκές είναι αυτή τη στιγμή να προτείνουμε ένα πακέτο κυρώσεων και ακατάλληλο μάλλον, όχι τόσο ανεπαρκές όσο ακατάλληλο. Το θέμα της μακροοικονομικής ισορροπίας ε, είναι κάτι καινοφανές σε σχέση με το παλιό πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης. Και ακριβώ επειδή πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο στοιχείο και στόχο έχει να διευρύνει ε, το πλαίσιο, γι' αυτό και θα πρέπει να είναι σωστό αυτό το πακέτο, το καινούριο πακέτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει δέσμευση, στενή δέσμευση στη διαδικασία από την αρχή, όπως προβλέπεται στη διαδικασία συναπόφαση και όχι μόνο στο σκέλος για τις κυρώσει, σε όλη τη συζήτηση, ώστε να καταλάβουμε τι ε, ζητούμε και τι, σε τι θα επιβάλλουμε κυρώσει. Εργαστήκαμε ε, σκληρά, άοκνα και ευχαριστώ την Προεδρία και την Επιτροπή για όλο το έργο και τη συνεργασία τη. Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη καταξουσιοδότηση πράξη και σε μια προσπάθεια συμβιβασμού ανταλλάξαμε τις κατεξουσιοδότηση πράξη προκειμένου να έχουμε ένα πλέγμα διατάξεων που είχε ως επίκεντρο την σφαιρική αντιμετώπιση Ευρώπης και όχι την κατακεδερματισμένη ανά χώρα με προκαταλήψεις για τις, για τις κυρώσεις. Κυρώσεις έχουμε ήδη αρκετές. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η περιπλοκότητα μια λειτουργία μια κοινή αγορά με κοινέ οριζόντιε πολιτικέ είναι τεράστια. Γι' αυτό το θέμα συμμετρία δεν είναι καθόλου ε, δευτερεύον. Βρίσκεται στο επίκεντρο τη κατάσταση και μα αυτά θα καταλάβουμε τι συμβαίνει και στην εσωτερική αγορά και στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να κρατήσουμε την ισορροπία που βρήκαμε με την Προεδρία. Και πραγματικά είναι απογοητευτικό που χάσαμε ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που κατέβαλαν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουμε την κοινή μας θέση και ευελπιστώ ότι με τις διαδικασίες που προσπαθούμε να κρατήσουμε θα συγκεντρώσουμε ακόμη, και, ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία για το πακέτο, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ένα σημαντικό σημείο στην έκθεση για την έλλειψη ισορροπίας, το θέμα της συμμετρίας συμμετρίας Αυτό δεν μπορούμε να το θυσιάσουμε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το συνεργάσιμο πνεύμα τους. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα λάθος βήματα. Γιατί τα λάθος βήματα δυστυχώς είναι πιο ορατά και πιο α, ε, έχουν προβληθεί περισσότερο από τα σωστά βήματα. Σωστά βήματα όμως είναι που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ο Κάρολ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την Ουγγρική Προεδρία για τις προσπάθειες ε, που μας έφεραν εδώ που βρισκόμαστε. Βέβαια η κατάσταση μπορούσε να είναι κάπως ευκολότερη, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό να δεχτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις πολιτικές διαφορές και ορισμένες από αυτές δεν μπορούν να επιληθούν παρά μόνο με την ψηφοφορία. Αλλά αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας. Ελίζα, μπράβο γιατί βρήκαμε κοινή θέση για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση μετά από πολλούς συμβιβασμούς, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό και θα ήθελα να διαβεβαιώσω την κυρία Φεραίρη ότι θα στηρίξουμε τη συμφωνία και την συμμετρία-συμμετρία γιατί είναι σωστή αυτή η προσέγγιση και ελπίζω να την κατανοήσει και το Συμβούλιο. Προσωπικά, όταν μιλούμε για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, λυπούμε που οι σοσιαλιστές δεν θα το υπερψηφίσουν και ταυτόχρονα υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μας και δεν νομίζω ότι μπορεί να την επιλύσει αυτή τη διαφορά οποιαδήποτε διαπραγμάτευση συμβαστική λύση. Δεν έχει καν νόημα να παρατείνουμε τη διαδικασία αυτή και χαίρομαι που η πλειοψηφία είναι υπέρ της ψηφοφορίας την Πέμπτη. Κάτι που ε, μεταθέτει την ευθύνη, το μεγαλύτερο τμήμα τη ευθύνη αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Ο κύριος Λάμπερτ είπε ότι ο τρόπος που ε, χειρίστηκαν το ζήτημα Γαλλία και Γερμανία δεν ήταν και πολύ επικοδομητικό. Το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πέμπτη και Παρασκευής έχει τεράστια ευθύνη για να εκτιμήσει την κατάσταση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δοθεί, να φανεί μία βούληση για συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ήταν κρίμα να λάβει το Συμβούλιο μια λάθος απόφαση. Νομίζω ότι η δική μας γραμμή είναι σωστή για να επιλύσουμε το πρόβλημα και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο Διέγκο. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός και εγώ Σάρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι και, και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω θερμά τους και ηγητές για τη δική μου έκθεση, αλλά να ευχαριστήσω και τα μέλη του Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής για τις ατέρμονες ώρες τριμερούς διαλόγου που είχαμε και μερικές φορές με μεγάλες διαφορές στις θέσεις μας. Οι γραμματείες και των τριών θεσμικών οργάνων και ιδιαίτερα η γραμματεία της Επιτροπής εργάστηκαν εργοδός και θα ήθελα να πω για, το δικό μου, για τη δική μου έκθεση ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι βρήκαμε έναν τρόπο λογικής εφαρμογής και για τον τρόπο, για τον χρόνο μείωση του δημόσιου χρέους και για το ρυθμό ε, μείωση του δημόσιου χρέου. Συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των παραγόντων. Συμφωνήσαμε. Τώρα για τη μεταβατική περίοδο για ορισμένες χώρες επίσης συμφωνήσαμε. Πέραν του διορθωτικού σκέλους θα ήθελα να επιμείνω και στην ανάγκη των ε, λύσεων που βρήκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, την ευφιέστερη εφαρμογή του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη, τον οικονομικό διάλογο, τα ευρωομόλογα, αλλά και το θέμα της συμμετρίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και απαραίτητο για να έχουμε μια Ευρώπη που θα αναπτύσσεται με λογικούς ρυθμούς. Και ελπίζω στην ψηφοφορία της Πέμπτης να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη πλειοψηφία ώστε να ενισχύσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η έκκλησή μου Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Πρέπει να πω στους βουλευτές πως και ε, ο Επίτροπος ε, και οι Υπουργοί ε, προσφέρθηκαν να παραστούν αλλά τους είπα πως οι βουλευτές θα είχαν ούτως ή άλλως πολλά να πούν από μόνοι τους και έτσι είναι πράγματι αλλά πρέπει να σου πω πως ήταν διατεθειμένοι να έρθουν ξέρω πως ε, υπάρχει θυμός για την ε, καθυστέρηση της τελικής ψηφοφορίας αλλά για να είμαι μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και ελπίζω το Συμβουλίο να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να πω πως η αναθεώρηση αυτής της ε, αντιστρόφου ειδικής πλειοψηφίας ε, δεν έχει φτάσει καν μέχρι την τη μέση, οπότε δεν πρέπει να τους εκπλήσει ότι το απορρίπτουμε. Το γεγονός ότι δεν επιτύχαμε συμφωνία αυτή την εβδομάδα δεν οφείλεται στην ε, συναπόφαση. Νομίζω ότι επιτύχαμε αρκετά πράγματα και νομίζω πως ένα σημαντικός παράγον ήταν η Ουγγρική Προεδρία και ο άντρα, ε, ο οποίος έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε να γίνει και Ζητώ συγγνώμη για το ότι σα κράτησα στην καρέκλα κολλημένους μέχρι τις 3 το πρωί, αλλά νομίζω πως εάν προωθήσαμε την τελική συμφωνία. Νομίζω αυτό οφείλεται και σε εσά. Αλλά βεβαίως ε, λογικό είναι όταν έχουμε τέτοιο πολιτικό ζήτημα να συνεχίζουμε να αναζητούμε συμφωνία και βεβαίως θα πρέπει να γίνει αυτό και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο μέσω του Συμβουλίου και διακυβερνητικών μέτρων. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε, γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε ευρεία πλειοψηφία για κάποια από τα ζητήματα αυτά στο Κοινοβούλιο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ακριβώς αυτή η ε, πλειοψηφία και η συμφωνία. Και θα έλεγα στο Συμβούλιο πως ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι μέσω της εμπλοκής του Κοινοβουλίου. Και άρα θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορία της ε, Πέμπτης. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ε, με καθυστέρηση 15 λεπτών θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με την Πόλα Ανκόξ, Πρωθυπουργό της Βερμούδας και Υπουργό Οικονομικών και ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Right, Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ησυχία. Έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και μετά έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον ε, Ούγκρο Υπουργό Οικονομικών, μετά από την ε, Πρωθυπουργό των Βερμούδων. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά όπως παρατηρήσατε είχαμε κάποια ε, σημαντικά ζητήματα ε, και καθυστερήσαμε λίγο. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θέλουμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε και δεν θα καθυστερήσω άλλο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα στους ε, κυρίες και κυρίους βουλευτές και τους προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι μοναδικό βεβαίως για Πρωθυπουργό και βουλευτή από το, τις Βερμούδες ε, να έχει την ευκαιρία να μιλάει ενώπιον σας. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί νομίζω πως ε, πραγματικά αυτό το οποίο έχει αξία είναι η ανταλλαγή απόψεων. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό να σημειώσουμε είναι πως βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την ευκαιρία να είμαστε ένα στρατηγικός εταίρος και βεβαίως υπάρχει και ειδική σχέση ε, είχα πάρα πολλές συναντήσεις αυτές τις μέρες. Ε, συναντήθηκα και με την Επιτροπή ΑΚΕ, τη Γραμματεία, με της ε, Επιτροπής Φορολογίας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και είναι σημαντικό το ότι έχουμε την ευκαιρία, ειδικά δεδομένων των όσων συμβαίνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πως είναι μια εβδομάδα μεγάλων αναδραχών με ενέργεια και δεδομένων των όσων συμβαίνουν εντός της Ευρώπης, αλλά νομίζω πως αποτελεί ευκαιρία και για εμάς να έχουμε έναν διάλογο. Και το λέω αυτό γιατί μόλις την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Ουάσιγκτον, εκεί πέρα το Κογκρέσο ασχολείται με το τι θα κάνει το ζήτημα της αύξησης της νομοθετικής οροφής ε, που υπάρχει στο χρέος, γιατί θέλουν να παραλύσουν οι ΙΠΑ. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν ζούμε τις επιπτώσεις της ύφεσης ε, που ήταν άνευ προηγουμένου τα τελευταία χρόνια και νομίζω πως ε, τα σχόλια τα οποία έκανε ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Γκάιτνερ τον είπα στις αρχές του μήνα όταν είπε πως ελπίζει ε, λόγω της σοβαρότερης εποπτείας που υπάρχει στις ΗΠΑ να μην υπάρχει πλέον ένα ρυθμιστικό αμπριτράζ και να διαλέγουν άλλες χώρες που ε, έχουν ε, έναν ε, μικρότερο βαθμό εποπτείας. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό και από πλευράς Βερμούδας παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά το ότι το ρυθμιστικό μας πλαίσιο πρέπει να είναι εύρωστο και να παίζει έναν προληπτικό ρόλο. Και η δουλειά που έχει κάνει η εποπτική αρχή της Βερμούδας και πρέπει βεβαίως να πω πως είναι και ο πρόεδρος της εδώ πέρα σήμερα καθώς και μέλη του προσωπικού του. Ε, αυτό γίνεται γιατί ως χώρα θεωρούμε πως είναι σημαντικό να έχουμε εύρος τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να συνειδητοποιούμε πως απαιτούνται συστημικές προσαρμογές. Από τη δική μας τη σκοπιά όσον αφορά το, το μέγεθός μας. Πριν από λίγες εβδομάδες φιλοξενήσαμε το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΣΑ. Γιατί, γιατί είμαστε στην αντιπροεδρία, αλλά σημαντικότερο είναι η εντύπωση που θέλουμε να δώσουμε για την δέσμευσή μας, την διαφάνεια και την συνεργασία. Όλοι στην διαβάρκα είμαστε και ο κόσμος είναι πραγματικά ένα χωριό που γίνεται όλο και πιο μικρό. Τα οικονομικά συστήματα μας είναι αλληλένδετα και αναγνωρίζουμε πως έχουμε τώρα μια ευκαιρία και πρέπει να είμαστε σαφείς και αποφασιστικοί στις δεσμεύσεις μας για το μέλλον. Η δε... Ο δε οίκος ή και ε, αξιολόγησης μας επένεσαν όσον αφορά την δέσμευσή μας για τη νομοθεσία περί φερικιότητας 2 ε, γιατί επιδείξαμε ξεκάθαρα πως δεν αστειευόμαστε και αναγνωρίζουμε την σημασία της αξιοπιστίας, της ακαιρεότητας και υγιών δομών και ενός γενικότερου πλαισίου ε, λειτουργίας και όσον αφορά ε, ολόκληρο το πλέγμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οπότε, θα έλεγα, ολοκληρώνοντας, πως εάν πρέπει ένα πράγμα να συγκρατήσετε για τις Βερμούδες είναι το εξής παρά το μικρό μας μέγεθος θεωρούμε εαυτόν γίγαντες και όχι ψήλους θα έλεγα όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας και της διαφάνειας. Και έχουμε 24 συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχει, όπως σας είπα, αυτό το σύστημα το εύρωστο και αξιόπιστο και τρίτο και τελευταίο, θα έλεγα, πως ε, ξέρετε, οι λέξεις ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη ισχύουν ακόμα και για ένα νησί το οποίο δεν είναι τόσο κοντά γεωγραφικά, αλλά ε, είναι κοντά όσον αφορά το ότι έχουμε κάποιες κοινέ Αρχέ λειτουργίας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο έχει πολλές προκλήσεις. Ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ήδη ζήτησε το λόγο ο Πίτερ Σκίνερ που ήταν και ο συγητής για το δεύτερο παγιάτο φερικιότητες. Οπότε φαντάζομαι ξέρεις πολλά για, τις Βερμούδες. Μακάρι να ήξερα πολύ περισσότερα. Πάντως, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την έλευσή σας εδώ και για την εκθέση των απόψεών σας. Παρά διπλωματική διπλωματικοί πάντως, γιατί συναντήθηκα με συναδέλφους σας και γνωρίζω ότι υπάρχουν λόγοι που ε, οι Βερμούδες αποφάσισαν να αυξήσουν το βαθμό διαφάνειας και να αλλάξουν τις διαδικασίες. Βέβαια πάντα οι κριτικοί λένε ότι θα μπορούσε κανείς να είναι πιο φιλόδοξος, αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι που θέσαμε ψηλά τον πύχη για τις περισσότερες χώρες και είστε από τις πρώτες χώρες, ανήκετε στην πρώτη ομάδα χωρών που ζητάτε ισοδυναμία. Μόνο οι, οι η Ιαπωνία και η Ελβετία είναι ε, σε τέτοια θέση. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντίληψη που έχουν πολλοί για το τι συμβαίνει offshore και πολλοί θεωρούν ότι δημιουργεί κίνδυνο για τις οικονομίες γιατί δεν εκφεύγουν οποιοδήποτε ελέγχο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για αυτό. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούτε περισσότερο τους Αμερικανούς ή τους Ευρωπαίους γιατί η γεωγραφική σας θέση ακριβώς ανάμεσα στους δύο σας δίνει αυτή την ε, ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά κάποια προϊόντα τέτοια οικονομικά και πολλοί Ευρωπαίοι θα φοβούνταν ε, τέτοια προϊόντα λόγω του κινδύνου ίσως που εμπεριέχουν. Αλλά φαντάζομαι ότι το έργο το... της χώρας σας είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να εγκομιάσω αυτά που συμβαίνουν εκεί και φαίνεται σταθερή η πρόοδο σα. Δεν ξέρω αν ε, υπάρχει κάτι από εμά που περιμένατε, γιατί αναφερθήκατε στην στρατηγική σχέση. Ε, σε αυτές τις διατηλαντικές σχέσεις τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί το θέμα αυτό των διατηλαντικών σχέσεων είναι ιδιαίτερα προσφυλές για μας, όπως ξέρετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σίγουρα είναι πολύ σχηδής ε, περίπλοκη και παρόλο που είμαι δικηγόρος θα προσπαθήσω να είμαι ε, συνοπτική στην απάντηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αντίληψης και της διχοτομίας μεταξύ offshore και onshore, οι Βερμούδες είναι ε, πολύ ειλικρινείς και ξεκάθαρη σταράτη στην προσέγγιση της. Δεν θέλουμε ε, να αποτρέψουμε τις χώρες που θέλουν να επενδύσουν. Θέλουμε να τις εξασφαλίσουμε ένα νομοθετικό, κανονιστικό και προληπτικό πλαίσιο ανεφροηγουμένου για να είναι πραγματικά ένας ασφαλής προορισμός. Και μάλιστα έχουμε ε, από τους αυστηρότερους οργανισμούς και ε, αρχές που μας αξιολόγησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαμε μια οργάνωση της ε, μεγάλη Βρετανίας και πριν από δύο εβδομάδες και μια αξιολόγηση της φερεγγιότητας και όταν μιλούμε για διαφάνεια και συνεργασία, δεν θέλω να πω ότι πριν από πολλά χρόνια οι Βερμούδες συμμετείχαν στον ε, πρότυπο κώδικα για την φορολογική διαφάνεια του ΟΣΑ. Θελήσαμε να πρωτοστατήσουμε και στη συμμετοχή αλλά και στην διαμόρφωση της καλύτερης της κατάστασης και να ε, αποδείξουμε ότι συμμετέχουμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Ό,τι αφορά την αξιοπιστία λοιπόν και τη δέσμευσή μας ε, είναι σαφής η πορεία μέχρι στιγμής των Βερμούδων. Σε ό,τι αφορά τις, ε, την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, είμαστε την πρώτη χώρα που μπήκε στο λευκό κατάλογο γιατί είναι σαφές ότι αν θέλουμε να είμαστε παγκόσμιος εταίρος και ε, ενεργός φορέας στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και να το αποδεικνύουμε αυτό σε όσους θέλουν να έχουν ε, εμπορικέ και οικονομικές συναλλαγές με τις Βερμούδες. Θα πρέπει να δείξουμε την καλή μας φήμη γιατί η αξιοπιστία και η καλή φήμη είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, ακόμη και με βάση τις αμερικανικές προδιαγραφές και τους ε, κανονισμούς για την πάταξη της λεύκανσης ε, χρήματος. Είμαστε από τις χώρες με το λιγότερο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή την ε, νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και από αυτήν την άποψη είμαστε ιδιαίτερα αξιόπιστοι. Οπότε το θέμα onshore και offshore. Μιλούμε με τις επιδόσεις μας Είχαμε την περασμένη εβδομάδα 200 εκπροσώπους από όλες τις χώρες ε, γιατί διοργανώσαμε το φόρουμ του ΟΣΑ. Αναλάβαμε την αντιπροεδρία του ΟΣΑ και το δείξαμε αυτό λοιπόν, δείξαμε την αξιοπιστία μας με τη, μέχρι τώρα μέτρα μας. Ό,τι αφορά το, τη φερεγγιότητα 2, ε, τις αντασφαλίσεις και τα οικονομικά. Πολύ συχνά όταν υπησερχόμαστε σε τέτοια θέματα, ε, γιατί μερικές φορές όταν μιλώ στο κοινοβούλιο για τα οικονομικά είναι πραγματικά ακούγονται πολύ αποκριφιστικά και τεχνικά. Δεν έχουν καμία σχέση με τα κοινωνικά για παράδειγμα. Όταν όμως μιλούμε για ε, διάφορες πράξεις όπως για τα captives και τα commercial reassurance δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Τα captives είναι ένα ειδικό προϊόν αφορούν ένα τμήμα των ασφαλίσεων, οπότε ο κίνδυνος για τους ψηφοφόρους, τους πελάτες είναι χαμηλότερος, γιατί έχουμε συγκρατήσει τον κίνδυνο. Τώρα, για τα κάπτυψη, του, τους εμπορικούς ασφαλιστές υπησέρχονται σε άλλη κατηγορία. Είναι πολύ πιο σημαντική και το είδαμε και από τη ρυθμιστική αρχή των Βερμούδων, ότι έχουμε ένα κανονιστικό σύστημα που στηρίζεται στις αρχές αλλά και λαμβάνει υπόψη και τον κίνδυνο. Και βλέπετε από την νομοθεσία μας ότι α, υψώνουμε όλο και περισσότερο τον πύχη, κάνουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους στην ανεξάρτητη αυτή ρυθμιστική αρχή και εγώ, Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εθνική Οικονομία, συζητούμε στο Κοινοβούλιο όλε τι νομοθετικέ προτάσει, ώστε να υπερκεράσουμε όλα τα εμπόδια. Είναι πολύ σημαντικό για όσου αξιολογούν τι Βερμούδε να αναγνωρίσουν τι διαφορέ μεταξύ των captives που δεν ενέχουν τόσο κίνδυνο και τις, ε, τα μέτρα για, τον ε, εμπορικό, για την εμπορική αντασφάλιση τις πολύ, τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Οπότε, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ο ρόλος των Βερμούδων ε, και το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται. Είχαμε 16 δις ετησίως και οι εισαγωγέ έχουν αυξηθεί από το 500 ε, εκατομμύρια σε 1,5 δις από το 2007. Το συνολικό εμπόριο Γερμανίας με τις Βερμούδες έχει αυξηθεί κατά 50% το εμπόριο υπηρεσιών και 100% εισαγωγής ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις Βερμούδες. Και νομίζω ότι η εμπειρογνωμοσύνη μας έγκυται στις ειδικευμένες, στα ειδικευμένα προϊόντα και ο κόσμος έρχεται σε εμά όχι για τις απλές δουλειές, αλλά για τις περίπλοκες ειδικευμένε, γιατί έχουμε και τα προσόντα, τις δεξιότητες και καινοτόμες γνώσεις που πληρούν και τις προδιαγραφές των πελατών αλλά και της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Οπότε από αυτήν την άποψη και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εποφελούνται από το μεγαλύτερο ανταγωνισμό και το χαμηλότερο κόστος. Και όταν πήγα στην Ουάσιγκτον αυτό το θέμα κυρίως επισήμανα. Γιατί μπορεί να λέω πόσο καταπληκτικοί είμαστε και πόσο υγιείς ε, είναι οι κανονισμοί μας και ποια είναι η ακεραιότητά μας και η καλή μας φήμη. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους πολιτικούς είναι γιατί ε, τους ενδιαφέρουν οι ψηφοφόροι τους, ε, η τοπική βάση, είναι πώς επηρεάζονται οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια, πώς καταπολεμάται η νομοποίηση παράνομων εσόδων ή πώς ε, θα προστατευτούμε από πλημμύρες, από τυφώνες κτλ. Και να μειωθεί φυσικά το κόστος και για τους τόπιους ε, καταναλωτές. Και αυτό είναι που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από τα τεχνικά περίπλοκα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση και σε τι προσβλέπουμε, θα ήθελα να σας δώσω ένα ε, σήμαντο παράδειγμα. Χθες, κάνοντας μια βόλτα και έχοντας συναντήσεις με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ρώτησα, γιατί ξέρω ότι όσα θα έχει ένα αποσπασμένο στη Βερμούδα ένα νέο γιατί υπάρχει μεγάλη, μεγάλος φόρτος εργασιών και όλες οι χώρες θέλουν έκθεση αλλά ακριβώ επειδή έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη θα αποσπάσουν κάποιον, θα στείλουν κάποιον ε, με κόστος της κυβέρνησης των Βερμούδων αλλά θα υποφεληθούμε και εμείς από αυτό γιατί μετά από ένα-δύο χρόνια θα έχουμε κάποιον που θα είναι σημείο επαφής ε, και θα έχει συγκεντρώσει και την δέουσα πείρα. Και μάλιστα Χθε που είχα συναντήσει με πολλούς ε, διευθυντές της επιτροπή, ρώτησα υπάρχει η δυνατότητα ή η προθυμία να έχουμε αποσπασμένους και από τη Βερμούδα εδώ, όχι με, δικό σας, ε, με δικά σα έξοδα. Θα τους χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση, εκτός και αν υπάρχουν βέβαια, αλλά γιατί ασκείται πολλές φορές επικρίσεις στις Βερμούδες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα εταιρική σχέση. απόσπασμένη υπάλληλοι από και προ τι Βερμούδε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, είναι σημαντικό και να αναφέρει τη Βερμούδα ω το χώρο του πρώτου κύματο αξιολογήσεων. Και ευκταίο φυσικά κάτι τέτοιο. Γιατί εμείς έχουμε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, έχουμε λάβει τα μέτρα και κάναμε ό,τι μπορούμε για να σεβαστούμε τι προδιαγραφέ και μάλιστα σε πολύ σύντομο διάστημα. Αυτό που θα ήθελα να σας ε, διαμηνήσω είναι ότι εσείς ως συνομοθέτες και ως ε, σχεδιαστές πολιτικής θα πρέπει να εξετάσετε το θέμα της ισοδυναμίας με το πακέτο Φεργκιώτα 2 και να μην ε, πληγεί η Βερμούδα, οι Βερμούδες να μην πληγούν λόγω, της λόγω των προσπαθειών και εξαιτία της επιμέλειάς της γιατί έδειξαν μεγάλη συνεργασία και έσπευσαν να τηρήσουν τις προδιαγραφές, να μην βρεθούν χαμένοι όμως εξαιτίας αυτής της επιμέλειας και να μην βρεθούν τιμωρημένοι εξαιτίας του ζήλους τους αυτού. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα νομίζω της στρατηγικής μας ε, εταιρική σχέσης. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική αυτή απάντηση. Φιλίπ, να ευχαριστούμε κυρία Πρωθυπουργέ που είστε εδώ σήμερα. Για να είμαι ειλικρινή, εγώ έχω πρόβλημα να αντιληφθώ γιατί οι εταιρείε, πολλέ εταιρείε και από την Ευρώπη, τη είπα, θένε να στήσουν ε, έδρα στη Βερμούδα. Ξέρω πως έχει το ωραίο καιρό βεβαίως. Μπορεί να έχετε και κάποια πύρα κτλ. αλλά εγώ θα έλεγα πως τέτοια πύρα μπορεί να βρεθεί και αλλού και σε τόσο πιστοδρομικές ε, υπήρους όπως η Ευρώπη ή η Βόρεια Αμερική. Οπότε, εάν έρχονται σε εσά. Ε, δεν είναι για λόγους αναπτυξιακής βοήθειας, μάλλον γιατί μεταφράζεται άμεσα σε κάτι σε χρηματικό όφελος. Και μπορείτε να το πείτε εσείς όπως θέλετε, αλλά αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι από πλευράς διαφάνειας οι ισολογισμοί στην χώρα σας ε, δεν δημοσιεύονται, η ιδιοκτησία των εταιριών δεν καταγράφεται δημοσίως, οι λεπτομέρειες της ιδιοκτησίας τίποτα, δεν θέλετε να ε, συμμετάσχετε στην οδηγία φορολόγησης ε, των καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εντάξει, μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ Βερμούδας και άλλων χωρών, εντάξει, ομολογουμένως δεν κάνετε τα χειρότερα, αλλά θα αρχίσω να σας ε, πιστεύω όταν ενταχθείτε στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές και εφαρμόσετε την Ευρωπαϊκή Οδηγία Φορολόγησης Καταθέσεων. Εάν λάβετε τέτοια βήματα, τότε θα σκεφτώ, ναι, αυτές οι κυρίες και οι κύριοι είναι σοβαροί αλλά ακόμα δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για την ερώτηση και το σχόλιο και προφανώς ε, θα διαφωνήσω και θα σας πω γιατί. Εγώ έγινα τέλη Οκτωβρίου πρωθυπουργός ε, της χώρας μου και μία από τις δηλώσεις που έκανα είναι πως δεν θα συνεχίσουν τα πράγματα ως συνήθως και πως οι Βερμούδες είναι ανοιχτές για να δεχτούν επιχειρήσεις. Και είναι σημαντικό, ε, μια που αναφερθήκατε στο ωραίο περιβάλλον της χώρας μας, νομίζω πως το 1970 οι Βερμούδες ήταν γνωστές για την ε, ροζ άμμο και τους ουρανούς και την ηρεμία, αλλά έχει αλλάξει πλέον το ποσοστό επιχειρήσεων και διακοπών και τώρα είμαστε γνωστοί για τις εγκαταστάσεις μας, ε, τις ικανότητές μας και την φήμη μας ως ε, μια χώρα που προσφέρονται χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και όπως σας είπα έχει μεταβληθεί αυτή η αναλογία σε σχέση με τον τουρισμό και όπως είπα και για το σχόλιο με τις ε, συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και για το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΩΣΑ, πως δεν τίθεται ζήτημα για το πόσο εύρωστο είναι το πλαίσιό μας και για τις πράξεις μας. Και θα σας έλεγα πως όσον αφορά την οδηγία περί αποταμιεύσεων. Η Βερμούδα δεν ήταν στον κατάλογο, αλλά έχουμε πει στις διαβουλεύσεις μας, στις συζητήσεις μας, πως πιστεύουμε στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών από τη δεκαετία του 80 με τις ΗΠΑ και ως αρμόδια αρχή όταν λαμβάνουμε αιτήματα οπωσδήποτε ανταποκρινόμαστε με εξαιρετικό τρόπο. Οπότε νομίζω πως η πιο πολύ σωστά σκεπτόμενοι άνθρωποι ε, βλέπουν ε, την καλή μας πίστη και πως το ότι είμαστε θα έλεγα συντονισμένοι και εμείς όσον αφορά την ακαιρεότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Αυτό προσελκύει τις επιχειρήσεις στη Βερμούδα. Η φήμη, η φήμη και η καλή μας φήμη. Και το ότι ξέρουν ότι δεν είμαστε κάπου πεταμένοι μόνο με πολλές τράπεζες, έχουμε τέσσερις τράπεζες και ε, οπωσδήποτε συμφωνούμε με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οπότε είμαι σίγουρη πως σε το χρόνο θα αλλάξετε άποψη. Αλλά ευχαριστώ για τα σχόλια σας. Ευχαριστώ Αστρίντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη, αλλά τα αγγλικά μου δεν είναι πια και τόσο καλά. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πρωθυπουργό των Βερμούδων που ήρθε στην Επιτροπή μας. Και θα ήθελα κυρίως να τη συγχαρώ. Να σας συγχαρώ κυρία μου για τον τρόπο με τον οποίο μας εξηγήσατε την προσπάθειά σας ε, ε, υπέρ της αξιοπιστίας, ε, της τιμιότητας της αξιοπιστίας ε, στις δημοσιονομικές αγορές. Και εγώ από μια μικρή χώρα έρχομαι, το Λουξεμβούργο, και οι μεγάλοι και, εμεί, εμείς υποκείμεθα από τους μεγάλους τις ίδιες κριτικές, διότι παρότι είμαστε μικροί ε, αναπτύσσουμε τη χρηματοπιστωτική μας αγορά και άλλους ε, οικονομικούς τομείς. Ορισμένοι μεγάλοι θεωρούν ότι οι μικροί δεν πρέπει να ανακατεύονται με τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σας καταλαβαίνω. Και θέλω να σας συγχαρώ και να σας πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και το ξέρω από την εμπειρία μου εδώ στο κοινοβούλιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πολεμάει κανείς ε, ε, κατά των παλαιών ε, προκαταλήψεων και όπως λέει και η παροιμία του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα και η τελευταία τοποθέτηση αποδεικνύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή διατυπώνονται αβάσιμες κρίσεις που δεν βασίζονται στα γεγονότα αλλά στις προκαταλήψεις. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα κράτη-μέλη, ε, τα ευρωπαϊκά κράτη θα πηγαίνανε στις Βερμούδες ε, να ανοίξουν μια επιχείρηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα label playing field. Level, συγγνώμη. Αμοιβαία δηλαδή και όταν άλλοι έρχονται να ανοίξουν ε, μια επιχείρηση στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αμοιβαίο σεβασμό των κανόνων. Τώρα για τα μέσα προσέλκυσης έχουμε λύσεις. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε διότι είναι συμβατές και σέβονται τους κανονισμούς. Πρέπει να αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα όπως έχουν για να είμαστε δηλαδή και ικανοποιητικοί όσον αφορά στα θέματα ρευστότητες. Κυρία μου, μπορούσα να μακρηγορήσω, αλλά νομίζω πως τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θέλω να σας πω πως η ηγεσία είναι το να κάνει κανείς το σωστό. Οι Βερμούδες θεωρούν αυτόν ηγέτη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οπωσδήποτε θεωρούν πως πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Γι' αυτό και έκανα το σχόλιο το ότι ελπίζω να μην τιμωρηθούμε ως ε, στο απολωλό πρόβατο. εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για τα... Thank you very much. You, you, Είστε τυχεροί, λέει η πρόεδρο. Ε, έχετε τους ε, τρεις ανθρώπους που προσπάθησαν να ζήσουν το, ζήτημα αυτών των captives στο πλαίσιο της οδηγίας ε, περί 2. Αν το λένε, ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας ε, στην Επιτροπή. Εσείς ε, θέσατε την ε, αρχή της στρατηγικής συνεργασίας, μιλήσατε για τις Βερμούδες και για τις χρησματοποιήσεις πιστοτικές τους υπηρεσίες. Εγώ θα ήθελα όμως να ρωτήσω για τη συνεργασία σχετικά με την εποπτεία. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Δηλαδή να υπάρχει εγγύηση ότι γίνεται η εποπτεία και της δίνεται και η απαραίτητη πληροφόρηση στις ευρωπαϊκές αρχές. Τώρα, δεύτερον, φορολογική συνεργασία. Υπάρχει βούληση για φορολογική συνεργασία η οποία να ευνοεί μια ανταλλαγή πληροφοριών και θα μπορούσαμε να έχουμε τις αντίστοιχες προδιαγραφές αυτής της παροχής πληροφοριών όπως έχουμε και στην Ευρώπη με τα κράτη-μέλη και θα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες πληροφόρησης country by country, χώρα προς χώρα Sir, thank you for Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δύο πτυχές ε, για το πρώτο ερώτημα που ήταν το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την ε, συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές. Τι πάνω πει ε, ανεξάρτητος. Ε, στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί είμαι και Υπουργός Οικονομικών, έχουμε την ανεξάρτητη εποπτική αρχή στην οποία δεν ανακατεύομαι ούτε εγώ ούτε η πολιτική. Ε, δεν ξέρω, μπορεί κάποιο να πει πως γι' αυτό ίσως εργάζονται τόσο καλά, αλλά αυτό το οποίο θα έλεγα είναι πως η νομισματική αρχή της Βερμούδας έχει συστήσει τα υποπτικά σώματα σε διεθνές επίπεδο και έρχονται σε επαφή με υποπτικές αρχές σε όλο τον κόσμο εν αναμονή της ε, φεργαιότητας 2 και ισοδυνάμων μέτρων, πρέπει να υπάρχει διάλογος ε, για τα λειτουργικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν απαραίτητες πληροφορίες για τις εταιρείε ε, που έχουν ε, σε ολόκληρο τον κόσμο για να υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο θηγατρικές για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών παγκοσμίω. Αυτό λοιπόν κάνουμε εμείς. Και μάλιστα ήμουν εδώ αυτή την εβδομάδα γιατί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα και ε, κράτους ε, με την ε, ρυθμιστική αρχή ήταν ε, και υπομορφή συμμετοχή μας σε διάλογο αυτή την εβδομάδα. Και ταυτόχρονα προσκαλέσαμε ρυθμιστικές αρχές από όλο τον κόσμο στις Βερμούδες πέρσι νομίζω κάπου, κάπου και Οκτώβριο-Νοέμβριο γιατί και πάλι η νομισματική αρχή της χώρας μας ε, φρόντισε γι' αυτό γιατί το θεωρεί σημαντικό. Λοιπόν, σε ένα πρωινό εργασίας που είχα σήμερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε πως ε, υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας και διάθεσης να δούμε και τη ρυθμιστική πλευρά για την δυνατότητα αποσπάσεων. Τίποτα δεν ορίστηκε συγκεκριμένα, αλλά τουλάχιστον δείχνει αυτό πως ε, δεν μένουμε στον τύπο ε, και να υπερτερεί ο τύπος της ουσίας. Θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι αμοιβέ ανταλλαγές πληροφοριών και η συνεργασία αυτή. Όσον αφορά τώρα τη φορολογική συνεργασία, όπως σας είπα, εμείς ήμασταν εξ αρχής στις προσπάθειες του ΟΣΑ όσον αφορά τον ηθικό το λεγόμενο κώδικα και ε, από, ξεκινώντας από χαμηλά έχουμε φτάσει στην κορυφή της λίστας και έχουμε πολλές ε, ε συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών προφών 24 και αυξάνονται. Αύριο θα πάω στο Λονδίνο όπου θα υπογράψω και εκεί πέρα συμφωνία και μετά θα ακολουθήσει συμφωνία ανάλογη με την Ινδονησία. Οπότε θα ε, είμαστε εμείς υπεύθυνη χώρα στο παγκόσμιο σκηνικό και οπωσδήποτε δεν θα κάνουμε βρωμοδουλειές. Δεν είναι αυτό το προφίλ μας, αν θέλετε. Ευχαριστώ, Θεόδωρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Πρωθυπουργό. για την, την, αποφαση, για την αξιοπιστία, την ομιμότητα κλπ. για όλες τις συνδιαλλαγές στις Βερμούδες και μεταξύ Βερμούδων και άλλων χωρών. Ο κύριος Λαμπερτέ έθεσε το θέμα των επιχειρηματιών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις Βερμούδες και όπου δεν δημοσιοποιείται το όνομά τους. Τι απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση, γιατί εγώ δεν την άκουσα. Είχε τεθεί μια ερώτηση για την καταχώρηση των εταιριών και το θέμα της προνομιακής ιδιοκτησίας. Ένα θέμα της νομοθεσίας μας που εμπίπτει και στην εντολή της ε, αρχής εποπτείας της ε, Βερμούδας είναι να γνωρίζει κανείς τον πελάτη για να αποφύγουμε την, ε, την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Και αυτό στα πλαίσια της καταπολέμησης λεύκας χρήματος. Είναι θέμα της προληπτικής ε, εξέτασης. Όταν φυσικά έχουμε μητρό επιχειρήσεων και έχουμε και την ε, ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που υπάρχει και το θέμα της προληπτικής αρνησικηρίας. Ελέγχεται η ταυτότητα αυτού που θέλει να ιδρύσει μια εταιρεία και γίνεται έλεγχος αξιοπιστίας του πελάτη και της καλής πίστης του υποψήφιου πελάτη. Ήδη λοιπόν έχουμε περιχαρακώσει όλα αυτά τα θέματα στις, ε, ε, στις ε, νομοθετικές μας Και υπάρχει και σχετική, σχετικός νόμος για τις εταιρείε. Και σε ό,τι αφορά την προνομιακή ιδιοκτησία, πρόσφατα υιοθετήσαμε μια νομοθετική πράξη στα πλαίσια της αξιολόγησης μεταξύ ισοτήμων Εκεί υιοθετούμε μία σταδιακή προσέγγιση και σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη νομοθεσία μας έχουμε και την προληπτική εξέταση, την προληπτική εποπτεία, υπάρχει το δυνατότητα βέτου και η εξέταση και η καταχώρηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στι φερμούδε. Φυσικά υπάρχει τέτοιο μητρό, ανοιχτό στο κοινό, μπορεί κανεί να το επισκεφτεί στι εργάσιμες ώρε. Και φυσικά μπορεί να βγάλει και αντίγραφα. Είμαστε διαφανείς και είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή η ανάγκη της διαφάνειας. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, Όποιο και είναι το ιστορικό μιας μικρής χώρας έξω από ένα ισχυρό οικονομικό μπλοκ, πολλές χώρες εντός του οικονομικού μπλοκ θα προσπαθούν, όπως ρώτησε και ο Φιλίπ, να εξηγήσει τι είναι αυτό το πονηρό ίσως που καθιστά τόσο δημοφιλή αυτή τη μικρή χώρα και έχει αναπτύξει τόσο μεγάλο, τόσο ισχυρό κλάδο. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν υπήρχε φορολογικός ανταγωνισμός υπήρχε κάποια διαφάνεια ή έλλειψη διαφάνειας τέλος πάντων. Πάντως, από τη στιγμή που οι χώρες του οικονομικού μπλοκ βλέπουν ή περιμένουν να, να δουν ότι οι μικρές αυτές χώρες συμμορφώνονται, περιμένουν ότι οι επιχειρήσεις θα φύγουν. Όταν εξακολουθούν να παραμένουν, οι χώρες υποπτεύονται ότι εξακολουθεί να παραμένει κάτι πονηρό σε αυτή τη χώρα που τις ελκύει. Βέβαια, κάποιες μικρέ χώρε έχουν και συγκριτικό αποτέλεσμα. Έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα μάλλον, γιατί έχουν πραγματογνωμοσύνη, έχουν γνώσεις, έχουν γίνει ανταγωνιστικέ με διαφάνεια και συμμορφωμένες προς τις γενικέ απαιτήσει και τις διεθνεί διατάξεις. Δεν ξέρω πώς μπορώ να διασκεδάσω κάποιες υπόνοιες χωρών ή υπηκών χωρών που θεωρούν ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, αν αυτό ρωτάτε. Πάντως έκανα ένα διαχωρισμό. Νομίζω ότι οι Βερμούδες είναι ένα, μια χώρα που έδειξε με μεγάλο πνεύμα συνεργασίας, διαφάνεια και συμμόρφωση. Το έχει αποδείξει αυτό. Κάτι που προβληματίζει πολλούς και το θεωρούν και παράδοξο είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί μια τόσο μικρή χώρα μπορεί να είναι ελκυστική για τους επενδυτές. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες μικρές χώρες ή για άλλες χώρες, ούτε θέλω να τις κατηγορήσω, αλλά αυτό που μπορώ να πω για μας είναι ότι μιλούμε για, ανεξάρ... για ανεξάρτητες ε, αξιολογήσεις. Έχουμε αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την έκθεση Food, και γνωρίζουμε με βάση αυτούς τους ανεξάρτητους ελέγχους και τις αξιολογήσεις ότι οι Βερμούδες έχουν, συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο που ακόμη και ο καθηγητής Κούμενς από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο είπαν ότι οι Βερμούδες εφαρμόζουν αυτό το cluster effect. Τι εννοεί ο καθηγητής λέγοντας το cluster effect, ότι υπήρξε μια συσσόρευση ταλέντου, δεξιότητας, εμπειρογνωμοσύνης, τεχνικών γνώσεων και σε ό,τι αφορά το επίπεδο και την εμβέλεια των ε, επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εκεί, αλλά και εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών. Οπότε έχουμε αξιόπιστες τράπεζες, Έχουμε δικηγόρους που θεωρούνται κορυφαίοι, έχουμε επιχειρήσεις ε, λογιστικού ελέγχου, επίσης ε, κορυφαίες. Οπότε δημιουργείται ένας πόλος έλξης, ε, γίνεται μαγνήτης η χώρα αυτή. Και ταυτόχρονα ήμασταν και καινοτόμοι στην προσέγγισή μας και τηρήσαμε και ένα πακέτο που είναι υγιές διασφαλίζει την καλή μας φήμη και περιλαμβάνει και προληπτική εποπτεία. Όλα αυτά τα στοιχεία ελκύουν τις επιχειρήσεις της Βερμούδας. Και ένα από τα βασικά μας χαρακτηριστικά είναι ότι εφαρμόζουμε και μεγάλη ταχύτητα. Μία επιχείρηση μπορεί εύκολα να μπει στην αγορά, γιατί από τη στιγμή που ξεπεράσει αυτόν τον προληπτικό έλεγχο και το δεν υποβληθεί βέτο, δεν ε, γύρουμε προς κόμματα. Μπορεί αμέσω να άρχισει να λειτουργεί μια επιχείρηση πολύ γρήγορα. Ταχύτητα είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Για να είναι κανεί ανταγωνιστικό, θα πρέπει να διευκολύνει τι επιχειρήσει να εγκαθίστανται και να ξεκινούν να λειτουργούν. Και από τη στιγμή που τηρούμε ένα σωστό πλαίσιο, που είναι προληπτικό, υγιές, ε, έχει καλή φήμη, ε, τηρεί του κανονισμού και τι διατάξει. και εξακολουθεί να διασφαλίζει την ε, θελκτικότητα των Βερμούδων ως βασικό πόλο χρηματοπιστωτικών ε, επιχειρήσεων, αυτό παραμείνει. Και εγώ προσπαθώ να έχω συναντήσει με επιχειρήσεις και πολλές φορές λένε ότι παρόλο που το κόστος μπορεί να μην είναι τόσο διαφορετικό από άλλες χώρες, αυτό που ενδιαφέρει στις Βερμούδες είναι η ποιότητα, η φήμη και η προσπελασιμότητα. Ε, μπορεί κανεί εύκολα να συναντήσει τον Υπουργό Μετανάστευση, Υπουργό Οικονομικών, Βερμούδε, να συναντήσει εκπροσώπου τη ρυθμιστική αρχή. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση με τι αρμόδιε αρχέ. Και εμεί ανταποκρινόμαστε και επίση έχουμε, έχουμε μεγάλη ποιότητα παροχή υπηρεσιών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν το συγκριτικό πλεονέκτημα των Βερμούδων. Και είμαστε άλλωστε μια χώρα που είναι πανέμορφη, το τοπίο είναι ωραίο και συμβάλλει σε αυτό σε μια επιπλέον τέρψη πέραν του οικονομικού ωφέλους και της ε, ελκυστικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως τελείωσαν εδώ οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ξέρω πως ε, κάποιοι βουλευτές όπως και εγώ θα συνεχίσουν το διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές σας. ειδικά στο πλαίσιο της ε, Φεργιότητας 2 και άλλων νομοθετημάτων για να βρούμε έναν τρόπο να βρεθεί κάτι ισοδύναμο. Καθώς μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ όσον αφορά τις προδιαγραφές, αλλά δεν πρέπει να δημιουργούμε ε, ένα φράχτη γύρω από την Ευρώπη και εμείς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και είμαι ότι θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, διάλειμμα 5 λεπτών για να δούμε το τι θα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια και θα προσπαθήσω να βρω και τον κύριο Υπουργό. Έχουμε τον Ούγκρο Υπουργό που θα έρθει. Uh, um, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω πως ε, δεν ξέρω, υπέγραψα εδώ πέρα να δώσω τα πρωτότοκα παιδιά μου. Εν πάση περιπτώσει, τα έγγραφα πρέπει να φύγουν. Λοιπόν, ορίζω τον ε, Ούγκρο Υπουργό Οικονομικών, Γιώργη Ματόλση, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και... Υπουργό Οικονομικών στην Ουγγαρία και χαίρομαι που καλωσορίζω και τον παλιό μας φίλο τον άντρε Κάρμεν και αναρωτιόμασταν τι, πώς επιζήσαμε χωρίς εσένα τις τελευταίες μέρες γιατί βεβαίω σε όλους αυτούς τους τριμερείς διαλόγους έχουμε συνηθίσει πλέον ο ένας στην παρέα του άλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή και αναμένουμε να μας πείτε και την δική σας την, άποψη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σάρων. Ο άντρε είναι, είναι μέλος εδώ της Λέσχης, της Επιτροπής Οικονομικών. Είμαστε υπερήφανοι και είμαστε υπερήφανοι για το ότι και εσείς τον δεχτήκατε. Να πω λοιπόν, κύριε και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Σάρων, αγαπητοί Σάρων, Είμαστε στις τελευταίες ημέρες της Ουγγρικής Προεδρίας, οπότε θα ήθελα να συνοψίσω τους στόχους και τα αποτελέσματα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας των τελευταίων σχεδόν έξι μηνών. Εάν ε, μου επιτρέπετε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για την εξαιρετική στρατηγική συνεργασία που είχαμε. Αποδείχθηκε κέριος ο ρόλος σας για την Ουγγρική Προεδρία, καθώς τις τελευταίες έξι εβδομάδες είχαμε εκτεταμένες ε, συναντήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς ε, διαλόγου. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, μας βοήθησε να εκπροσωπήσουμε έτσι, μια κοινή προσέγγιση στο ΕΚΟΦΗΝ. Οπότε, θεωρώ πως επιτύχαμε πολλά με τη βοήθειά σας. Δεύτερον, να πω πως ε, βασικός ε, στόχος σημερινής μας συνάντησης δεν είναι να ληφθούν αποφάσεις. Έχουμε ήδη λάβει δηλαδή, τις αποφάσεις χτες ε, εμείς στο Συμβούλιο Υπουργών και εσείς θα λάβετε τις δικές σας αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίω όλοι οι πολιτικοί, ενώ οι πρωθυπουργοί μας δηλαδή, θα λάβουν και αυτοί τις αποφάσεις τους. Αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή λήψης των αποφάσεων. Είναι η στιγμή όμως να σκεφτούμε τη στρατηγική μας ε, συνεργασία του τελευταίους μήνες να ξαναδούμε την ε, συνεργασία μας και να σας ε, ξανακούσουμε στο τέλος της προεδρίας μας. Να συνεχίσω λέγοντας πως κατά την Ουγγρική Προεδρία εστιάσαμε σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα βεβαίως ήμασταν εντός του Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κοφίν βεβαίως και είχαμε δύο ιστορικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Να πω πως οι δύο αυτές ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ιστορικές ε, εξελίξεις καθώς όσον αφορά το πακέτο αυτό διακυβέρνησης αποτελεί ένα πρώτο βήμα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και επίσης το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένα ιστορικό εγχείρημα γιατί είναι μέρος της συνολικής απάντησης στην κρίση και είναι και πάλι η πρώτη φορά που ε, καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές και νομίζω πως ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες γιατί τα επιτύχαμε και τα δύο από πλευρά Συμβουλίου Οπότε επιτύχαμε μια γενική συμφωνία στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και χτες εγκρίναμε όλες τις συστάσεις της ε, Κομισιόν, οπότε πλέον είναι συστάσεις ε, του Συμβουλίου για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή και το πρόγραμμα σταθερότητας και το πρόγραμμα σύγκλησης. Οπότε έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο σημαντικά εγχειρήματα και αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως ιστορικά βήματα ελπίζουμε προς σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως εκτός του Συμβουλίου, πέρα από αυτό, έπρεπε να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Ε, είχαμε την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ε, Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, είχαμε την Ελλάδα, τους G20, αλλά έπρεπε να ασχοληθούμε πρώτα με το πρώτο ε, ζήτημα, δηλαδή τα στρατηγικά βήματα για το μελλοντικό πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και βεβαίως φαίνεται πως τα πράγματα πήγαιναν όπως συνήθως, αλλά καταφέραμε να περάσουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οπότε αυτοί οι τρεις φάκελοι θα έρθουν μαζί με άλλους τις επόμενες μέρες σε εσά. και μαζί με τα υπόλοιπα δηλαδή το πακέτο όπως ανέφερα, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Οδηγία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Να πω επίσης πώς βεβαίως Το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης είναι το πιο σημαντικό ε, καθήκον που έχουμε να ολοκληρώσουμε, αλλά σε αυτή τη στιγμή η τελική απόφαση είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου. Προσωπικά θεωρώ πως η απάντηση που δώσαμε στην κρίση και η πρόληψη μελλοντικών κρίσεων ε, δεν θα είναι επαρκής ε, λύση χωρίς το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Το εξαπλώτο το λεγόμενο. Ήταν λοιπόν κοινή προσπάθεια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και είμαι περήφανος για την καλή συνεργασία που είχαμε. Και εξ και της Ουγγρικής Προεδρίας και του Άντρας να σας ευχαριστήσω για την στρατηγική αυτή συνεργασία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό για την Προεδρία μας. Πρέπει να τονίσω πως ε, μετά τη θέση ενισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας αυτά είναι η πρώτη φορά που Συμβούλιο και Κοινοβούλιο υιοθετούν νομοθεσία με τη διαδικασία της συναπόφασης στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ιστορική αυτή τη διαδικασία. Γιατί ήταν η πρώτη φορά, όπως σας είπα, που έγινε με συναπόφαση και πρέπει να τονίσω πως η εμπειρία της Ευρώπης ε, από τη συνεργασία των διεθνικών οργάνων είναι πάρα πολύ θετική. Ως Προεδρεύον του Συμβουλίου πρέπει να παραδεχτώ πως κατά τη γνώμη μου οι τροπολογίες ε, του Κοινοβουλίου βελτίωσαν αισθητά το κείμενο. Οπότε, εξ ονόματος της Ουκρικής Προεδρίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, τροπολογίες. Πώς ήταν, 2079? Πόλες, κάπου τόσες. Ξέρετε, ως, ως πρόεδρος του, του ΕΚΟΦΗΝ πρέπει να, να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό το νούμερο δηλαδή πρέπει να το ξέρω απ' έξω. Τέλος. Όσον αφορά το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης θα ήθελα να πω πως ο στόχος ε, και Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι ο ίδιος, δηλαδή να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και της Ευρωζώνης και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών σοκ. Είναι ο δικός σας ο στόχος και ο στόχος ε, του Συμβουλίου επίσης, οπότε είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον και είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για οριστικοποίηση του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης. Οπότε, το Συμβούλιο συμφώνησε χτες σε ένα συμβασμό, όπως ξέρετε, το οποίο το αποστήλαμε στο Κοινοβούλιο, το οριστικό κείμενο δηλαδή χτες. Ελπίζουμε οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν μετά από 70 ώρες ε, τριμερούς διαλόγου 70, ε, και περισσότερες μου φάνηκαν ειδικά, ειδικά και σε σας σαν θα φάνηκαν περισσότερες και στα μέλη της ε, Επιτροπής σας Ο Επίτροπος δεν είναι εδώ λοιπόν να κάνω μια παρατήρηση λοιπόν για τον ρόλο του. Η Κομισιόν ήταν ειλικρινής διαμεσολαβητής και παρά το που σιάζει ο κύριος Ολυρέν θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το εξαιρετικό του έργο. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις απετέλεσε και αυτό ένα θεμέλιο λίθο του έργου μας και νομίζω πως το πρώτο αυτό εξάμεινο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές. Χτες το Συμβούλιο ενέκρινε συστάσεις αναχώρα και για την Ευρωζώνη. Ήταν η πρώτη φορά, ξεκίνησε λοιπόν η όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θεωρούμε όλες οι στάσεις χρήσιμες για τη βελτίωση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Οι συστάσεις αυτές βεβαίως ακολούθησαν την αξιολόγηση της Κομισιόν για τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα αυτό αργότερα αυτή την εβδομάδα. Τέλος. Τέλος, να πω πως πολλά οικονομικά ζητήματα, το μιλάμε για το ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα ολοκληρώσαμε και καταφέραμε συνολικά να προωθήσουμε πέντε φακέλους και θα υποβάλουμε δύο φακέλους σε εσά που σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας μας μαζί με το Κοινοβούλιο. δηλαδή το ένα αφορά τους ε, χρηματοοικονομικούς ομίλους και το άλλο τη μεταφορά μετρητών σε ευρώ. Είχαμε και τις προτάσεις λοιπόν για τις υπηρεσίες στο Συμβούλιο και τα σοβαρά επιτεύγματα όσον αφορά και την κάλυψη ακάλυπτων πωλήσεων, ε, ασφαλίστερων κινδύνου, τη γενική προσέγγιση για την οδηγία Εγγύσεων καταθέσεων και το Όπω Όπως ξέρετε λοιπόν, Σάρων, αγαπητοί συνάλφοι, θα έλεγα πως ήταν αρκετά ευχάριστη η συνεργασία μας όλους αυτούς τους μήνες στο πλαίσιο της Ευρώπης. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν. Αυτό είναι τριμερής διάλογος, η δημοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο στις χώρες μας. Ξέρετε είμαι βουλευτής στην Ουγγαρία και είμαι υπέρ του δημοκρατικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεργασία και ελπίζω το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ολοκληρώσει το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης στις ερχόμενες μέρες και εβδομάδες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, and... Σας ευχαριστούμε και για τα ευγενικά σας λόγια. Ήταν όντως uh, ταραχώδες το κλίμα μερικές φορές, αλλά όπως είπατε κι εσείς, Είχαμε διαπραγματεύσεις για θέματα πολύ σημαντικό και πέραν της οικονομικής διακυβέρνηση και μερικά καταφέραμε θέματα να τα φέρουμε σε αίσιο πέρα. σε μερικά κολλήσαμε λίγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αμφισβητείται, υπονομεύετε το έργο της Ουγγρική Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι βάλετε πραγματικά όλοι σας την ψυχή στις συζητήσεις, ιδιαίτερα για το πακέτο της μακροοικονομικής διακυβέρνησης και χωρίς τη δική σας επιμέλεια και ζήλο δεν θα βρισκόμασταν στο σημείο που βρεθήκαμε. Και έχουμε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε λίγο καιρό ακόμη πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και ελπίζω να βρούμε τελική λύση. Ο Ζαν Πολ. Κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Υπουργέ, Δύο παρατηρήσεις. Μία ειλικρινή και μία πιο μακροσκελή. Η ειλικρινή μου παρατήρηση είναι για να σας ευχαριστήσω για την ποιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας και να σας πω πόσο εκτιμήσαμε την ε, ε, διαθεσιμότητά σας προς εμάς. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με την Ουγγρική Προεδρία και η Ουγγρική Προεδρία πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της ικανοποιημένο για τη δουλειά της. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα της φιλικής ειλικρίνειας. Δεύτερο όμως που θα μακρηγορήσω είναι ότι δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας για την τωρινή κατάσταση. Εμείς έχουμε δύο σοβαρά πράγματα που παραμένουν ανοιχτά ακόμα το ζήτημα της Ελλάδας και ακόμη και αν το Κοινοβούλιο δεν ερωτήθηκε άμεσα για το θέμα το οποίο παραμένει διακυβερνητικό ή διμερές αυτό είναι κρίμα διότι η κατάσταση έχει ιδιαίτερη επίπτωση στα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά στις επιπτώσεις του ευρώ έστω και αν πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το πρόβλημα του ευρώ, είναι το πρόβλημα του χρέους της Ελλάδας. Και κρίμα που τον Μάιο του 2010 συνδέσαμε το πρόβλημα της Ελλάδας με το ευρώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Από τη μια το πρόβλημα Ελλάδα και από την άλλη το πρόβλημα ευρώ. Για την οικονομική διακυβέρνηση τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα διότι το Κοινοβούλιο εξέφρασε ζητούμενα, το Συμβούλιο αντέδρασε, σας ευχαριστούμε, αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά δύσκολα σημεία τα οποία διαταράσσουν το προχώρημα αυτών των δύο ζητουμένων. Το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να λυθεί σύντομα διότι παίζεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έστω και αν δεν συνδέεται άμεσα παίζεται και η αξιοπιστία για την προσπάθεια που γίνεται υπέρ της Ελλάδος. Τι παίζεται εδώ. Η ικανότητα των κρατών μελών να είναι από τη μια μεριά αλληλέγγυη και από την άλλη συντονισμένη στις οικονομικές πολιτικές. Όλοι το ξέρουν και το λένε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα και 17 και 27 διαφορετικές οικονομίες αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανασύρουμε τις επιπτώσεις της κρίσης τις οποίες δεν θέλαμε να ανασύρουμε πριν από την κρίση για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Αυτό πρέπει να λυθεί σήμερα. Δεύτερο, νομίζω ότι υπάρχει άγνοια των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ κοινοβουλίων και κρατών μελών. Για πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ως ένα εθνικό κοινοβούλιο στο οποίο μπορεί κανείς να δίνει οδηγίες και όπου έχουμε μία πλειοψηφία η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται στις ε, διατάξεις που δίνει το Συμβούλιο. Βέβαια αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαλύσει την κυβέρνηση, πράγμα που γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ειδικό σχεσιακό πρόβλημα το οποίο λύνεται μέσα από τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας μονομερός να καθορίζει τη θέση του. Σε ορισμένα σημεία όμως αυτή η συζήτηση δεν είναι πάντοτε σαφής και για να είμαι ρεαλιστής φοβούμε προσωπική άποψη είναι ότι χάνουμε πολύ χρόνο να συζητούμε γύρω από σημεία τα οποία δεν έχουν καμία πρακτική επίπτωση. Η πρόληψη δεν μπλέκεται διότι στο εγγύς μέλλον θα βρισκόμαστε σε φάση διόρθωσης, οπότε οι κανόνες για τη διόρθωση θα πρέπει να εφαρμόζονται και απ' την άλλη επίσης φοβούμε ότι αν προκύψει μια πραγματική κρίση, τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση δεν θα τα ψάξουμε μέσα από νομικίστικες ε, και δύσκολες διατάξεις αλλά θα κοιτάξουμε στα γρήγορα να το λύνουμε ψάχνοντας αλλού. Ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία για την εξαιρετική της δουλειά, αλλά έχω τις αμφιβολίες μου και τη θλίψη μου διότι έχουμε εδώ την ευρωπαϊκή προσπάθεια όπως επίσης και την θέση του κοινοβουλίου που εμπλέκονται και δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρουν όλα αυτά οι πολίτες μας. Επιμηκύνεται συνέχεια ο κατάλογος των αγορετών. Θα ακούσουμε τρεις ερωτήσεις και μετά θα ακούσουμε τι απαντήσει από το Συμβούλιο. Πρέπει να φύγει Κορίν, γιατί είναι η σειρά σου. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Προεδρεύοντα, για την παρουσία σας, εδώ κατά το εξάμεινο της Ουγγρικής Προεδρίας και ευχαριστούμε θερμά για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλατε και προσπαθήσατε να γεφυρώσετε με κάθε μέσο τις διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στο Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε καταθέτοντας 2.000 τροπολογίες, τις μειώσαμε σε 700 και βρέθηκαν στα χέρια του Άντερ Σκάρμαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι είναι μείζον επίτευγμα το γεγονός ότι την προηγουμένη εβδομάδα καταφέραμε να συμφωνήσουμε σχεδόν σε όλα τα ζητήματα. Μερικές φορές είναι αδύνατον ε, ταυτόχρονα να λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες. Αυτό που κάνουμε τώρα με το να θέτουμε σε ψηφοφορία αυτό το πακέτο είναι για να διευκρινίσουμε τη σημασία της πρόοδου που υλοποιήσαμε. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που είπε ο Ζαν Πολ Τεράστια ευθύνη φέρουμε όλοι μας και δεδομένη της ελληνικής κρίσης είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό πακέτο που θα μπορέσουμε να το θεωρήσουμε ως ε, στέρη βάση για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση και ταυτόχρονα να επιστρέψουμε στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχολησιμότητας για τους πολίτες μας. Έχω με δύο θέματα πολύ ευαίσθητα πολιτικά επιτάπητος και ελπίζω ότι με τις κοινέ μας προσπάθειες θα κατορθώσουμε να βρούμε λύση η διαδικασία που ακολουθεί το Κοινοβούλιο δείχνει ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τις θέσεις μας, να προσπίσουμε τις απόψεις μας, αλλά είμαστε ταυτόχρονα ανοιχτοί και σε επίτευξη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τα μέχρι τώρα σας επιδεύματα και πρόοδο και ελπίζω να ξεπεράσουμε τα εναπομείναντα εμπόδια τις υπόλοιπε εβδομάδες που μας έμειναν πριν το τέλος της Προεδρίας. Και εγώ θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω σήμερα για την ε, παρουσία σας και να σας ευχαριστήσω και για τη δουλειά σας κατά την Προεδρία. Η Ουγγρική Προεδρία ασκήθηκε για πρώτη φορά και για πρώτη φορά επίσης ε, έθεσε εγκινήσει τους μηχανισμούς ε, για την συναπόφαση σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έπαιξε η Προεδρία σας σημαντικό ρόλο σε αυτά τα τρία σημεία. Τα άλλα θεσμικά όργανα ανέπτυξαν θεσμικό σκεπτικό σχετικά. Ο κύριος ε, Τρισέ ε, ανέφερε την θέση του και μίλησε επίσης για μεγαλύτερη θεσμική συνεργασία και εμείς θα θέλαμε μεγαλύτερη θεσμική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Θα ήθελα να ξέρω αν μεταξύ ΕΚΟΦΗΝ και των άλλων οικονομικών υπουργείων μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα για το ελληνικό ζήτημα ε, εγώ νομίζω ότι δεν μιλάμε σωστά όταν λέμε ελληνική κρίση. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή κρίση, μια κρίση της Ευρωζώνης και πάνω παραπάνω από την οικονομική κρίση είναι πολιτική κρίση. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει εμείς εδώ να κρίνουμε είναι η καθυστέρηση και η έλλειψη απαντήσεων που οξύνουν το πρόβλημα. Εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Μιλήσαμε σήμερα για διακυβέρνηση τον ε, Μάρτιο εργάζεστε ακόμα στο ΕΚΟΦΗΝ γι' αυτό, αλλά χρειάζεται να έχετε μεγαλύτερη ελαστικότητα να συμφωνήσετε με το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είναι μια ισορροπημένη λύση, διότι αλλιώ θα είναι μια ψευτολύση. Η ισορροπημένη λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης ε, που μέσα από τα πλαίσια των προπτικών σύγκλησης και αυτό για να διασφαλιστεί και η αξιοπιστία μας προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη δουλειά σας. Θα ήθελα όμως ε, να ξέρω τι γίνεται με τα ε, ασφάλιστρα, με, με τα ασφάλιστρα κινδύνου και με το κυρίαρχο χρέος. Θέλω να ξέρω πώς έχουν οριμάσει τα κείμενα και θα ήθελα να ξέρω αν θα μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία τους επόμενους Uh, uh, Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ κύριε Προεδρεύοντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τα ευγενικά σας λόγια προς την Ουγγρική Προεδρία. Είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε και τη βοήθεια και την υποστήριξή σας και την είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Κάτι που μας βοήθησε όλους. Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη στιγμή διακυβεύεται. Γιατί η κρίση εξακολουθεί να σοβεί, αυτό είναι σίγουρο, δεν έχουμε ξεφύγει από την κρίση και η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, η καιρή είναι χαλεπή έχουμε κίνδυνο δημόσιου χρέους στην ε, νότια πλευρά της Ένωσης. Έχουμε την κατάσταση αυτή στην Ευρωζώνη και ταυτόχρονα το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης για το μέλλον. Τουλάχιστον ένα από αυτά τα εκρεμή ζητήματα θα πρέπει να τα διαθετήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε φυσικά να επιλύσουμε εντάχει την ελληνική κρίση, οπότε θα πρέπει να επιλύσουμε να διαλέξουμε την άλλη εκκρεμότητα και εκείνη να διευθετήσουμε. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχετε και εκεί απόλυτο δίκιο. Και οι δύο. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ ότι η κρίση είναι πολιτική. Και με δύο λόγια πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τον επόμενο μήνα. Γιατί εύκολες λύσεις για την ελληνική κρίση δεν υπάρχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κορίν για τα ευγενικά της λόγια και εγώ πιστεύω ότι ελάχιστα απέχουμε από την τελική συμφωνία. 99,9%, 98% ε, δεν ξέρω. Πάντως είμαστε πολύ κοντά στην υλοποίηση της τελικής συμφωνίας. Και η Ευρώπη χρειάζεται αυτή την τελική συμφωνία. Αυτό είναι σίγουρο και αναμφισβήτητο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο και από άποψη ε, διεθνών αγορών. Χρειαζόμαστε μια επιτυχία και ίσως η επιτυχία μας ε, είναι αυτό το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει για να υλοποιήσουμε το στόχο, το στόχο μας να κάνουμε και την, να διανύσουμε και το τελική ευθεία. Θα ήθελα επίσης να σας πω σε φορά την τελευταία ερώτηση ότι η πρώτη μου εντύπωση από τη συνεργασία Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν θετική. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε τα θεσμικά όργανα μεταξύ μας. Και μπορεί να μην είναι τόσο προφανής ε, η συνεργασία, αλλά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα. Αυτή ήταν η αρχική μου εντύπωση και εξακολουθεί να ισχύει ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και παρόλο που μερικές φορές είναι αργή και χρονοβόρα αυτή η διαδικασία, μερικές φορές ακαθόδης και δύσκολη, μερικές φορές δεν μας επιτρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά παρόλα αυτά λειτουργεί η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και συμφωνώ μαζί σας 100% ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε μία πολιτική κρίση με δημοσιονομικά μέσα, γιατί η κρίση είναι πολιτική και βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι θέμα που ξεφεύγει από την Ουγγρική Προεδρία. Εμείς επικεντρωθήκαμε στα καθήκοντά μας στο Συμβούλιο και οι χώρες Ευρωζώνης ασχολούνται με την ελληνική κατάσταση. Και τέλος, ό,τι αφορά το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, θα ήθελα να πω ότι εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο. Βέβαια είμαι εκφύσεως αισιόδοξο άνθρωπος και είμαι αισιόδοξο ότι θα καταλήξουμε στη σε συμφωνία γιατί είμαστε και υποχρονική πίεση μας πιέζουν για κάποια λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης το χρειαζόμαστε διακαώς. Είναι επιτακτική ανάγκη και για το μέλλον της Ευρωζώνης, αλλά και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δώσω το λόγο εδώ στον συνάδελφο για να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ και πάλι θερμά για τα ευγενικά σας σχόλια για την Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω πρώτα απ' όλα για, τους, ε, για το χρηματοοικονομικό κανονισμό και μετά για την οικονομική διακυβέρνηση. Για τον κανονισμό. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό κομμάτι της συνολικής αυτής απάντησης. Είχαμε την οικονομική κρίση, τραπεζική κρίση πρόσφατα, όχι μόνο την κρίση του δημοσίου χρέους. Σημαντικό είναι να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα και να εφαρμόσουμε καλύτερη ρύθμιση στον τομέα αυτών. Θα θυμάστε πως στην αποκορύφωμα της κρίσης είχαμε ακάλυπτες ε, πωλήσει ε, και την ανταλλαγή αυτών των ε, credit default swaps και είχαμε αυτή την, έχουμε αυτή τη νέα προσέγγιση τώρα ε, στο Συμβούλιο και έχουμε προχωρήσει αρκετά για να επιτύχουμε μια συμφωνία στο σχετικό κανονισμό και με το Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επίσης γνωρίζουμε πως το 2008 Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν ήταν εναρμονισμένες οι εγγυήσεις των καταθέσεων. Τα λεφτά πήγαιναν από τη μια χώρα στην άλλη και προσπαθούσε ο κόσμος να βρει παραθυράκια στο σύστημα. Τώρα έχουμε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που εναρμονίζει αυτό το πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτείται προχρηματοδότηση των ταμείων εγγύησης καταθέσεων για πρώτη φορά στην Ευρώπη και ελπίζω πως με την εντολή αυτή η Πολωνική Προεδρία να μπορέσει να συμφωνήσει μαζί σας και επίσης είναι επίσης σημαντικό δίδαγμα της κρίσης να μειωθεί ο κίνδυνος αντισυμβαλωμένου. Να υπενθυμίσω τι συνέβη μετά τη χρεοκοπία της, ε, των Lehman Brothers. Έχουμε λοιπόν μια νέα ριζοσπαστική λύση τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα το ΕΜΙΡ είναι μια συνολική ε, ρύθμιση της κατάστασης. Στους τελευταίους έξι μήνες επιτύχαμε λοιπόν τεράστια πρόοδο ε, όσον αφορά το φάκελο αυτό εντός του Συμβουλίου και χτες οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια πολιτική συζήτηση για τα υπόλοιπα ζητήματα και ελπίζουμε η Προεδρία του Συμβουλίου να είναι έτοιμη να ξεκινήσει ε, διάλογο με το Κοινοβούλιο και κάτι άλλο ακόμα που δεν σχετίζεται τόσο πολύ με την κρίση αλλά είναι πολύ σημαντικό για τους πελάτες. Ε, το λαό της Ευρώπης είναι ο νέος κανονισμός ε, ευρωπαϊκών πληρωμών. Έχουμε πάλι, όπως σας είπα, ένα γενικό πλαίσιο και έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις και ελπίζω με τον κανονισμό να υποφεληθεί ο λαός από αυτό το πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Τέλος, μία παρατήρηση για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Θα έχω την ευκαιρία να πω και κάποια λόγια στην ε, Ολομέλεια. Αυτό βλέπουμε στο Συμβούλιο. Πώς το τωρινό κείμενο, επί το έχουμε σχεδόν συμφωνήσει θα έλεγα, είναι πολύ καλύτερο και πολύ ψηλότερης ποιότητας από ε, το αρχικό. Συμφωνήσαμε λοιπόν να δεχτούμε τέτοια σημαντικά ζητήματα όπως η κωδικοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα μπορώ να σας πω πως ε, έχουμε καταλήξει σε κάτι σωστό. Στην αρχή φοβόμασταν να μπει αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στον κανονισμό Επίσης εκτιμώ πάρα πολύ την ιδέα του οικονομικού διαλόγου για τη βελτίωση της διαφάνειας ε, και της λογοδοσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Συμβούλιο χτες υποστήριξε την συμβιβαστική μας πρόταση για να μπουν και μεμονωμένα κράτη-μέλη. Επίσης θεωρώ πως η εισαγωγή των ε, τοκοφόρων ε, καταθέσεων στο πλαίσιο των μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνεί με τις αρχές που είχαν συμφωνηθεί στο Συμβούλιο και πιο πριν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πως θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις νωρίτερα αλλά προοδευτικά. Θεωρώ πως αναβαθμίσαμε επίσης την ποιότητα του πίνακα βαθμολογίας και το σχέδιο, το σχεδιασμό του. Τώρα έχουμε αυτή την διπλή προσέγγιση που αντικατοπτρίζει πολύ περισσότερο το τι μπορεί να περιμένει κανείς από τα αναλυτικά αυτά εργαλεία στο μηχανισμό αυτό επιτήρησης αλλά επίσης είχαμε και πάρα πολύ καλό συμβασμό όσον αφορά την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υιοθέτηση του πίνακα βαθμολογίας και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός το να υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης για ευρωαξιόγραφα, να μείνει ανοιχτή η πόρτα. Ξέρετε πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σχολιάσουμε, αλλά πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η πόρτα, να μελετήσουμε την πιθανότητα και τέλος θεωρώ πως ήταν τεράστιο επίτευγμα το ότι μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για την αναθεώρηση της αντίστροφης ειδική πλειοψηφία στις μακροοικονομικές ανισορροπίες σε δύο περιπτώσεις. Συμφώνησε επίσης χτες το Συμβούλιο να γίνει ρητή αναφορά στη ρήτρα αναθεώρηση στο προληπτικό σκέλος όσον αφορά την αντιστραμμένη ειδική πλειοψηφία και αυτό δεν είναι βεβαίως ε, άνευ ε, συνεπειών γιατί αποφασίστηκε να διευκρινιστεί και να επεκταθεί η δήλωση συμμόρφωσης οπότε επιπλέον τώρα υπάρχει σαφής ε, δήλωση που είναι συμμόρφωσης ή επεξήγησης και πρέπει να γίνεται δημόσια κάθε φορά σε κάθε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν ακολουθεί τη σύσταση της Κομισιόν αλλά και το πεδίο εφαρμογή επεκτάθηκε χθε, γιατί τώρα δεν καλύπτει μόνο συστάσεις αλλά και προτάσεις της Κομισιόν. Δύο σημαντικά βήματα για να ενισχύσουμε την προσέγγιση αυτή, συμμόρφωσης ή εξήγησης και ταυτόχρονα έχουμε περίτρα αναθεώρησης που σημαίνει πως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εάν δεν λειτουργήσει αυτή η προσέγγιση, τότε υπάρχει σαφή ανάγκη αναθεόρηση, τη ε, διαδικασία ε, λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο τη συμφόλου σταθερότητα και ταυτοχρονα εχουμε περιτρα αναθεωρησης που σημαινει πως ειναι ξεκαθαρα τα πραγματα εαν δεν λειτουργησει αυτη η προσεγγιση τοτε υπαρχει σαφης αναγκη αναθεωρησης της διαδικασιας ληψη αποφασεων στο πλαισιο της συμφωνου σταθεροτητας και αναπτυξης chosen earlier and now strengthened further. Γιατί βεβαίως είναι σαφές πως ο τρόπος λειτουργία που είχαμε μέχρι τώρα δεν λειτουργήσε. I'm hurrying you along because we've got three more members. Ας βιαστούμε λίγο γιατί ζήτησαν ακόμη το λόγο ο κύριος Χουντής, ο κύριος Μαργκάγιο και ο κύριος Λάγκεν. Θα τους ακούσουμε και τους τρεις μαζί και μετά θα ακούσουμε τον Υπουργό. Πρόεδρε, Πράγματι πρέπει να βιαστούμε. Ο χρόνος για αναλυτική συζήτηση έχει περάσει. Άλλωστε τελειώνει η Ουγγρική Προεδρία. Χαίρομαι που είναι ο πρόεδρος Εντάξει, υπάρχει μετάφραση. Ναι, λέω, επειδή τελειώνει και η Ουγγρική Προεδρία, αλλά τελειώνει και ο χρόνος της συνεδρίας, θα είμαι σύντομος. Ε, χαίρομαι που είναι μαζί μας ε, έχω πολλά ερωτήματα κύριε Υπουργέ και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι αφήσατε κενά στη σημερινή παρουσίαση αλλά στο γεγονός όπως θα ξέρετε ότι το τελευταίο εξάμενο και στο εξάμενο της δικής σας Προεδρίας δυστυχώς από την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αφαιρεθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας ευθύνη. Υπάρχει ακόμα μια ασάφεια τι θα γίνει από αυτού. Δεν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συζητήσουμε, πέρα από τις γραπτές ερωτήσεις, σε θέματα που μας απασχολούσαν και δεν νομίζω πως είναι δική σας ευθύνη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτήματα, δεν θα σας κουράσω γρήγορα. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας σας υπευλήθη από την Ελλάδα που έχει αυτά τα προβλήματα, Έτοιμα να ενεργοποιηθεί το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Αν είσαστε πρόχειρος. Δεύτερο, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα παρακαλούσα την προσοχή σας και αν έχετε κάποια απάντηση. Από όσο γνωρίζω η χώρα σας κάποια στιγμή ήρθε σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να πάρει ένα σχετικό δάνειο. Αν αυτή τη συμφωνία που κάνατε τη θεωρήσατε διεθνή συμφωνία, αυτή είναι η ερώτηση, τότε σας ερωτώ κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας του ΕΚΟΦΗΝ αναρωτηθήκατε αν η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα οικονομικά της Ένωσης, στους μηχανισμούς στήριξης στην Ευρωζώνη είναι σύνομη με τις συνθήκες. Αποφάσισε ποτέ το Συμβούλιο για αυτή τη Διεθνή Συμφωνία των Οργάνων της Ένωσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί δεν αποφάσισε ή δεν συναποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Και τέλος, ε, χάρηκα κύριε Υπουργέ ε, με το γεγονός ότι είστε εκλεγμένος. Αύριο εύχομαι να τα καταφέρετε πολύ καλά μόνο ως Υπουργό Οικονομικών αλλά και ως Βουλευτής. Η ερώτηση λοιπόν έχει τον εξής χαρακτήρα και αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πώς θα αισθανόσαστε ως βουλευτής του Ουγγρικού Κοινοβουλίου όταν μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν θα έχετε πολλά περιθώρια έως ελάχιστα να διαμορφώσετε και να προγραμματίσετε μια οικονομική πολιτική που να απαντά στις ανάγκες του ουγγρικού λαού αλλά θα είσαστε υποχρεωμένος κάτω από τη συνεχή εποπτεία και νουθεσία της Κομισιόν και των συνεχών εποπτικών ελέγχων ουσιαστικά να βάλετε την υπογραφή σας σε προαποφασισμένα πράγματα. Σταματώ εδώ γιατί ε, να μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την, για την παρουσία σας. Δεν υπάρχουν άστοχες ερωτήσεις, άστοχες απαντήσεις υπάρχουν. Ο Όσκαρ Βάιλ το έλεγε αυτό. Όλοι συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν μια ενιαία νομισματική ζώνη, δεν υπήρχε συντονισμός στις οικονομίες Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, διαπιστώσαμε ότι η νομισματική ένωση με, χωρίς πολιτική ένωση μοιάζει πολύ σαν, ένα, σαν τίγρης φυτοφάγος. Ο Τρισέ έχει άλλη θέση, ο Γιούνκερ, ο Τρεμόντι είναι υπέρ των ευρωομολόγων. Πώς θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην πολιτική ένωση όποια και να είναι αυτά τα εμπόδια γιατί το βασικό είναι να ξέρει κανείς την πορεία και μετά ξέροντας την πορεία μπορεί να εντοπίσει τα εμπόδια. Ναι, σύντομο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα η Γκρική Προεδρία νομίζω έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Και μια που είναι μέλος μιας ε, τρόικας. Ε, πρέπει να ολοκληρωθούν ε, όλοι οι φάκελοι μέχρι τις 30 του μηνός. Μπορεί να τα δώσει Πολωνούς. Μια χαρά θα είναι. Δεύτερον, ο Έλληνας συνάδελφος που μίλησε από την Κομμουνιστική Ομάδα θέλω να διαφωνήσω. Δεν είναι το βασικό θέμα ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, εδώ πέρα. Αυτό το κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια, όχι εμείς. Εμείς ελέγχουμε την Κομισιόν, όχι το Συμβούλιο και είμαστε συνομοθέτες. Οπότε ο κύριος Υπουργό δεν χρειάζεται να αιτιολογεί εδώ πέρα το τι κάνει το Συμβούλιο για πτυχές που άπτονται της εθνικής αρμοδιότητας, αλλά Έχω αμφιβολίες για το εάν είναι διατεθειμένο να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα το Συμβούλιο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ως συνομοθέτες. Εάν δούμε το πακέτο αυτό της οικονομικής διακυβέρνησης βλέπουμε πως πάντα το ΕΚΟΦΗΝ ήταν αυτό που δεν μπορούσε να συμφωνήσει και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και ήθελε να αποδυναμώσει την Κομισιόν. Πάντα το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ήταν αυτό και τώρα έχουμε μία αυτόματη διαδικασία την οποία πάλι απορρίπτουν. Ε, πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα εδώ πέρα. Και δεύτερον, και θέλω να τελειώσω εδώ πέρα, η ρύθμιση παραγόγων. Το Συμβούλιο υπό την Προεδρία σας τρεις φορές άλλαξε το πεδίο εφαρμογή. Όπως είχε προταθεί τα over the counter, μετά για όλα τα παράγωγα, μετά ξανά over the counter και τώρα όλα. Ε, εμείς ε, τηρούσαμε την πρόταση της Κομισιόν και τον G20 δεν κατάλαβα πως ε, επί Ουγγρικής Προεδρίας διαρκώς άλλαζε η κατάσταση. Ίσως μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Right, we'll lose uh, interpretation. Σε τρία λεπτά δεν θα έχουμε πια διερμηνία. Οπότε αν συνεχίσουμε θα συνεχίσουμε μόνο σε μία γλώσσα Γι' αυτό παρακαλώ να είστε και εσείς σύντομος, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Χουντή, η ελληνική λύση, η κρίση, το ελληνικό δράμα, η ελληνική τραγωδία δεν ήταν στο πρόγραμμα του ΕΚΟΦΗΝ γιατί το Eurogroup είναι αρμόδιο για την διαθέτηση αυτής της κρίσης. Ό,τι αφορά την Ουγγρική Βουλή, οι Ουγγροί κατάφεραν να αλλάξουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαμαρτυρηθήκαμε ε, για κάποιες συστάσεις και ειδικά αντιταχθήκαμε στη διατύπωση ενός ε, γράφου που στήριζε αυτές τις συστάσεις και τελικά η Επιτροπή άλλαξε ένα μεγάλο τμήμα του κειμένου. Αυτά ως προ την αρμοδιότητα του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, που ήταν Εθνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Μαργάγιο, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν νοείται φορολογική, δημοσιονομική, νομισματική ένωση από μόνη της, ξεχωριστά. Είναι σαν τη Γαλλία τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Αλλά χρειάστηκαν 200 χρόνια για να καταλήξουμε σε αυτή την ενιαία χώρα που αποκαλούμε Γαλλία. Δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε και εμείς 200 χρόνια, δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια πολυτέλεια χρονική. Πάντως σίγουρα η διαδικασία είναι πολύ αργή. Είναι μια πολύ χρονοφόρα διαδικασία για να καταλήξουμε σε μια πραγματικά ενοποιημένη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χρειαζόμαστε και δημοσιονομική και νομισματική ένωση και πολιτική ένωση και ευρωομόλογα και κάποια άλλα μέσα για να χειριστούμε τις κρίσεις. Και η κρίση είναι ακριβώς που μας ε, ενθαρρύνει και μας ε, οθεί να ενισχύσουμε όσο γίνεται την Ένωση. Έχουμε και λατινικό ρητό που μας το δείχνει αυτό και η κρίση είναι μεγάλη απόδειξη. Και εγώ, εν συντομία, για το θέμα των παραγόγων, το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συρρυκνώθηκε στα παράγωγα OTC, over the counter, και δεν κάλυπτε τα παράγωγα που ανταλλάσσονται στο χρηματιστήριο. Πάντως, ως ειδικό δεν βλέπω για ποιο λόγο τα, ο κίνδυνος είναι διαφορετικός στις δύο περιπτώσεις over the counter και αυτά του χρηματιστηρίου. Πάντως, ε, η Βελική Προεδρία προσπάθησε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή και να καλύψει και κάποια άλλα παράγωγα. Πάντως ήταν σαφές ότι τα κράτη-μέλη έχουν διστάμενες απόψεις. Προσπαθήσαμε να Ασχοληθούμε το θέμα και χάσαμε κάποιους μήνες προσπαθώντας να διαχωρίσουμε το θέμα του πεδίου εφαρμογής ε, σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με τις υποχρεώσεις αναφοράς, τις απαιτήσει διαφοράς, συμψηφισμού ή εκαθάριση μάλλον και της ε, ανοιχτής και δίκαιης πρόσβασης και ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση μεταξύ των ε, κρατών με αυτές τις βάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την πρωινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το απόγευμα στις 3 προβλέπεται συζήτηση με ένα μόνο θέμα, την Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση, έκθεση Hackmark. Ελπίζω κάποιοι να παραμείνετε και για την απογευματινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ θερμά την Ουγγρική Προεδρία και ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε για όλο σας το έργο. Ευχαριστούμε και εμείς. Thank you very much.